Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Ο κύριος Μπουζέκ έχει μια σημαντική συνάντηση και θα καθυστερήσει λίγο και μου ζήτησε να αναλάβω εγώ στη θέση του. Πρώτο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, μια έγκριση τη ημερήσιας διάταξης, την έχετε στου φακέλους σας και θα ήθελα επίσης να σα ενημερώσω ότι τα σημεία 12 και 13 έχουν αλλάξει σειρά. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή. Υπάρχει παρατήρηση για την ημερήσια διάταξη, όχι από ό,τι βλέπω. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο θέμα, έγκριση των πρακτικών της ε, προηγούμενης συνεδρίασης. Ε, τα πρακτικά περιλαμβάνονται και αυτά στους φακέλους. Πρόκειται για τις συνεδριάσεις 14 και 20 Απριλίου. Υπάρχουν σχόλια για τα πρακτικά. Αν ναι, όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα συζητήσουμε την κατεύθυνση προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και ε, θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή, τον Μάρεκ ε, Γκρόμπατσιφ από την Ευρώπη των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών να μας παρουσιάσει την έκθεσή του και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε τους κοιόδης εισηγητές. Μετά τους κοιόδης εισηγητές ε, θα μιλήσει ε, ο κύριος Μπίλεν ε, από την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κύριε Γκρόμπατσεκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσση, γλώσσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ξεκίνησαν την ε, εργασία πάνω στο θέμα της Ευρωπαϊκής ε, Ενεργειακής Ένωσης κάτι το οποίο βεβαίως απαιτεί εσωτερική συνεργασία και θα διασφαλίσει την ασφάλεια την ενεργειακή για τους ε, συμπολίτες μας. Η έκθεση αυτή βασίζεται και στις ε, προηγούμενες εκθέσεις, είναι το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Ε, και επίσης βασίζεται στους κανονισμούς περί αερίου του ορίζοντα 2020. Προς τα εκεί πηγαίνουμε λοιπόν. Και πρέπει να πούμε πως 60% το αερίου το εισάγουμε και 90% του αργού πετρελαίου. Ένα δισεκατομμύριο την ημέρα δηλαδή για ενέργεια ξοδεύουμε. Πρόκειται για το Υπάρχει για πολύ υψηλό κόστος και είμαι στη μεγαλύτερη αγορά ενέργειας του κόσμου και αυτό βεβαίως αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Πάρα πολλά κράτη-μέλη είναι πλήρως εξαρτημένα από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Άλλα κράτη-μέλη εξαρτώνται από την Βόρεια Αφρική ε, οι πηγές αυτές λοιπόν της ενέργειας είναι ασταθείς και άρα πρέπει να βρούμε άλλες σταθερότερες ε, χώρες οι οποίες θα αντισταθμίσουν τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στην αγορά. Για τις τιμές τώρα. Οι τιμές στην Ευρώπη είναι υψηλότερες από ό,τι στις είπα. και από την Κίνα και την Ινδία. Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι δύο ή και τέσσερις φορές υψηλότερες σε κάποια κράτη-μέλη ή και παραπάνω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξάρτησης από έναν και μόνο προμηθευτή. Οι τιμές ε, καταναλωτή δε, οι τελικές τιμές μετά τους φόρους ε, αυξήθηκαν ε, κατά 5% το 2012-2013. Τώρα, για τη σημερινή μας ε, στρατηγική. Αυτή πρέπει να συμφωνεί με την συνθήκη που αναφέρει ξεκάθαρα πως ε, το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών, οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται εκεί. Αυτή είναι μια γενική αρχή την οποία πρέπει να σεβαστούμε. πότε. Μιλάμε για το ότι θα πρέπει να έχουμε διάφορες πηγές ε, Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις, να κατασκευαστούν διασυνδέσεις και αγωγή. Προφανώς, βεβαίως έχοντας κατά νου την ε, σχετική νομοθεσία. Η Κομισιόν λοιπόν τι ρόλο παίζει εδώ πέρα. Η Κομισιόν συντονίζει σε περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε οι λύσεις να είναι αποδεκτές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και τελικά να φροντίσει να υπάρχουν δυνατότητες ε, αντίδρασης σε περιπτώσεις ανάγκης. Τώρα, το μέσα αυτό αφορά τις υποδομές στην ε, ανάπτυξη αυτών διασυνοριακών, αυτών διασυνδέσεων. Άλλος ένας τομέας ε, που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι τα ζητήματα τα ε, συμβατικά. Οι συμβάσεις αυτές είναι ένα μεγάλο παραθυράκι όσον αφορά δηλαδή την ε, κατάργηση κάποιων καταχρηστικών ρήτρων που έχουν επιβληθεί από τρίτες χώρες, ε, ειδικά στα κράτη-μέλη που εξαρτώνται πλήρως από έναν και μόνο προμηθευτή. Ο ρόλος λοιπόν της Κομισιόν πρέπει να είναι δημιουργικός, να στηρίξει τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία θα ήθελαν να ε, μπουν σε τέτοιες διαπραγματεύσεις και αυτό θα πρέπει να είναι βεβαίως σε συμφωνία με τους κανονισμούς που διέπουν ε, την εσωτερική αγορά και αυτά τα οποία ορίζει ο ΠΟΕ και αναφέρομαι εδώ πέρα στις ε, ευαίσθητες ε, πληροφορίες, τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν μας απασχολούν. Οπότε όλο, όλος αυτός, όλο αυτό το θέμα παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να φροντίσουμε όλες αυτές οι συμβάσεις ε, να είναι διάφανες και αυτό απαιτεί την συμμετοχή της Κομισιόν στις ε, διαπραγματεύσεις εξ ονόματος των κρατών μελών εκείνων που θα ήθελαν να είναι παρόντα στις ε, διαπραγματεύσεις και άρα έχουμε έναν ολόκληρο κατάλογο διατάξεων ακριβώς για να αποφύγουμε τέτοιες ε, καταχρηστικές ρήτρε. στις συμβάσεις εκείνες οι οποίες ε, είναι θέμα αντικείμενο αξιολόγησης στα κράτη-μέλη. Και προφανώς βεβαίως θα πρέπει να ενοποιηθούν ε, και να τυποποιηθούν αυτές οι συμβάσεις, αλλά αυτό είναι και θέμα θέλησης ε, των κρατών μελών. Δεν είναι ανάγκη να δημοσιευτούν οι λεπτομέρειες, αλλά κάποια σημεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για να τα ξέρει το κοινό. Ναι, υπάρχει συμμεταχείριση των ε, κρατών μελών. Τώρα, όσον αφορά την διαφοροποίηση των ε, πηγών ε, ενέργειας, που είναι ο στόχος μας βεβαίως. πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τις ΙΠΑ. Ε, ε, ανταγωνίζονται τα κράτη-μέλη με τις ΗΠΑ και πρέπει να διατηρήσουμε βεβαίω και ένα επίπεδο ζωής ανάλογο. Οπότε οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση κάποιας πηγής ενέργειας. Ε, το μείγμα αυτό το ενεργειακό πρέπει να περιέχει και συμβατικές και ανανεώσιμες ε, και ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να, νικεί. Πρέπει να υπάρχουν και οι τρεις πυλώνες για να δημιουργηθεί η Ενεργειακή Ένωση για να έχουμε μια σταθερή και αξιόπιστη παροχή ενέργειας. κάποιες πηγές ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά οπωσδήποτε θα δούμε το τι θα γίνει με τη συμφωνία TTIP και την εξαγωγή LNG και αργού πετρελαίου από τη ΣΥΠΑ, όπου μάλλον η κατάσταση θα αλλάξει. Και βεβαίως το θέμα είναι και το σχιστολιθικό αέριο στην Λατινική Αμερική και με συγχωρείτε αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά έχετε μιλήσει πάρα πολύ ώρα. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλα δύο ζητήματα, αν μου επιτρέπετε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δύο λεπτά και το πολύ. Για την εσωτερική αγορά αναφέρθηκα ήδη ε, και θα πρέπει όπως είπαμε να είναι η λύση η οποία θα βρεθεί αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε και το θέμα της ε, αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε νέες λύσεις και να γίνει κάποια εξοικονόμηση όσον αφορά την ε, χρήση στα νοικοκυριά και αναφέρομαι βέβαια και στον τομέα των κατασκευών. Αλλά να μην είμαστε υπερβολικοί. για να μην ε, προδιαγράψουμε τα πάντα από τώρα. Πρέπει να υπάρξει κάποιος βαθμός διαπερατότητας ε, από την θερμότητα και κάποιες άλλες λύσεις ε, βεβαίως ε, τεχνολογικές θα προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες. Τέλος, χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Να αναφερθώ και σε αυτό. Το θέμα αυτό δεν ε, συμβιβάζεται τόσο πολύ με την ουδετερότητα απέναντι στις πηγές ενέργειας. Θα μπορούσε να προκαλέσει αποβιομηχανοποίηση και μια διαρροή των ε, ρηπογόνων ε, βιομηχανιών και βεβαίως να προκαλέσει ανεργία. Η Κομισιόν τώρα λέει πως το πακέτο αυτό θα καταλήξει στην κατάσταση στην οποία κάποιες κοινωνικές ομάδες δεν θα μπορούν να πληρώσουν ε, το λογαριασμό για να έχουν ενέργεια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση έχει στόχο να μειώσει τις τιμές κατά 20%. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αρχή του 20 20 να μειωθούν δηλαδή οι εκπομπές κατά 20% και τα ορυκτά καύσιμα αλλά πρέπει να φροντίσουμε να αυξηθεί και το ποστό της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να φτάσει στο 20%. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολιτικές ομάδες τώρα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τον κύριο Γιούλη. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ τον κύριο Κρόπατσικ για την πολύ σκληρή δουλειά. Μέσα σε το σύντομο διάστημα μπορούσε να μα παρουσιάσει το πρώτο σκαρίφημα τη έκθεσή του για να μπορέσουμε να συστήσουμε ήδη κάποιε συγκεκριμένε προτάσει. Η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να είναι σχετικά ε, κενή, ε, κενοφανή έννοια, αλλά είναι τα ζητήματά τη γνωστά ήδη και τα έχουμε συζητήσει ω στόχου στην Επιτροπή μα εδώ και πολλά χρόνια και ως εκ τούτου πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία ε, είναι ακόμα προ συζήτηση. Θα ήθελα ιδιαίτερα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο να υπογραμμίσω τα θέματα στα οποία συμφωνούμε, υπεραδείγματι την εξορρόπηση των κύριων ε, πυλώνων ε, τη ενέργεια, την ανταγωνιστικότητα δηλαδή, την ασφάλεια στι προμήθειε και την αηφορία ή βιωσιμότητα. Ξεκινώ με τη σειρά λοιπόν. Πρώτον, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον με στασιμότητα και με ανεργία πρέπει να δοθεί έμφαση ιδιαίτερα στην βιομηχανική ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υποστηριχθεί η δημιουργία θέσεων εργασία, η εξασφάλιση χαμηλών τιμών ενέργεια στον καταναλωτή είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, για να εξασφαλίσουμε λοιπόν του στόχου σε, έναν, ε, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, απώλεια πόρων άνθρακα. Επίση, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι υποδομέ για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Ε, ορυκτά καύσιμα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα έχουν μεν μειωμένο αλλά συνεχή ακόμη ρόλο και παρουσία στην οικονομία μας. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερα ταχθεί πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής με μια ε, επιλογή για την οικονομία με χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα, χαμηλή συμμετοχή στα ποσοστά άνθρακα. Επομένως, αντί να επικεντρωνόμαστε στην ε, ε, στα ορυκτά καύσιμα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια οικονομία με λιγότερη συμμετοχή του άνθρακα στο μείγμα, με φιλόδοξα σχέδια αλλά και τις τα κατάλληλα κίνητρα, ιδιαίτερα ε, για να καλυφθεί από το ποσοστό αυτό το 40% της ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική λοιπόν για τη θερμότητα και επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε και για την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την ανάπτυξη. Πιστεύω επίσης ότι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία είναι, σε σχέση με τις κυβερνήσει των κρατών μελών, είναι να μπορέσουν τα κράτη-μέλη πλήρω να υλοποιήσουν την νομοθεσία και κυρίω το τρίτο πακέτο για την ενέργεια. Λίγα λόγια τώρα για τη συγκεκριμένη πρόταση εν ώψη των ανωτέρων. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ε, βιωσιμότητα, τα στοιχεία αυτά δηλαδή που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα στο έγγραφο του συναδέλφου. Ο στόχος ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της μείωσης της εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας μας προβληματίζει κάπως. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο στόχο που θα αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση της χονδρικής ε, και των τιμών εισαγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Τον εισηγητή δεν έχω άλλο χρόνο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τζανονάτο, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Γκρόμπατσιτς, για το έργο του παρά το γεγονός ότι η πρώτη εντύπωση που μας δόθηκε από την ε, ανάγνωση ανακοίνωσής του είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών που ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της και ε, τις σκέψεις του εισηγητή. Απομακρυνόμαστε από μια τοποθέτηση η οποία βαθμιδών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Επιτροπή μας είχε αρχίσει να εδραιώνεται θα ήθελα να σας πω με ποια σημεία διαφωνώ ιδιαιτέρως, αν και συμφωνώ στο τμήμα που αφορά ε, τη συμπτωματολογία. Όσον αφορά τα συμπτώματα συμφωνούμε. Ως προς τη θεραπεία για το πώς ε, θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα οι διαφορές μας είναι αρκετές. Καταρχάς ε, ο εισηγητής αλλάζει τη δομή των πέντε βασικών πυλώνων που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεχνάμε τελείως την ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Παραγνωρίζουμε ή σχεδόν ε, παραγνωρίζουμε το θέμα της εναρμόνισης. Δίνουμε νέα διάσταση στο όλο ζήτημα της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας και πολλά άλλα θέματα είναι προβληματικά και πηγαίνουν σε διαφορετική κατάσταση, ε, κατεύθυνση συγγνώμη, από αυτήν που είχαμε καθορίσει εμείς στο κοινοβούλιο μας, κυρίως από τα όσα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έκανε και πολύ μεγάλα βήματα προς τη ζωστή κατεύθυνση. Ελπίζω να μπορούμε να έχουμε κάποια βελτίωση και να μην έχουμε πιστοδρόμηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πραγματικά ελπίζω ότι τις διάφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία σύγκληση η οποία αφενός θα έχει ως εφαλτήριο αυτό το οποίο επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα αναπτύξει σιγά σιγά τα θέματα με βάση τις ε, γραμμές που έχουν ε, σύν χρόνο καθιερωθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σταθώ σε μία που είναι πολύ ουσιαστική για μένα. Εμείς θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα με ολοκληρωμένη διακυβέρνηση της ενέργειας. Δεν θέλουμε να καθορίσουμε κάτι που είναι ένα σύνολο συμφωνιών μεταξύ κρατών και κάθε χώρα να είναι αυτόνομη ε, στο σπίτι της. Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες θα δίνουν κοινέ κατευθυντήριες γραμμές, χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα έχουν ενιαίες αρχές για τη διακυβέρνηση της ενέργειας και πρέπει να έχουμε και σαφείς ιδέες για τους πέντε πυλώνες που αποδεικνύονται. Σίγουρα η ασφάλεια, σίγουρα το χαμηλό κόστος της ενέργειας που θα πρέπει να υπάρχει και στην Ευρώπη. Ε, σίγουρα όλο αυτό το τμήμα που συνδέεται και αυτό είναι ουσιαστικό, δεν θα πρέπει να το λησμονούμε ε, στις εκπομπές αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τις οποίες συνεισφέρουμε και θα πρέπει εμείς να μειώσουμε προκειμένου να μειώσουμε και την υπερθέρμανση του πλανήτη και υπάρχουν και θέματα για τα οποία έχουμε εκφράσει άποψη σε διάφορα ψηφίσματα ε, της χαμηλής χρήσης άνθρακα, ε, την ε, ενεργειακή απόδοση των συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια ε, και φυσικά όλα όσα πηγαίνουν, επαναλαμβάνω, προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ φυσικά θα ήθελα να συζητήσω και με όλους τους συναδέλφους, αλλά βεβαίως και με τον εισηγητή, για να καταλήξουμε σε κάποια κοινή θέση. Δεν μπορώ να μην δηλώσω ότι αυτή τη στιγμή πόρο απέχουμε από συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερσεν, εξονόμητος στο Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε στο σχέδιο αυτό. Θα ήθελα ιδιαίτερως να υπογραμμίσω κάποιες κύριες πτυχές που θέλουμε εμείς να μελετήσουμε περισσότερο, να καταθέσουμε τροπολογίε και περαιτέρω να επεξεργαστούμε. Για την διακυβέρνηση στο σχέδιο αυτό πολύ σωστά υπογραμμίζεται η σημασία τη ανάπτυξη μια πραγματική μια γνήσία Ευρωπαϊκή ενιαία αγορά για την ενέργεια έτσι ώστε να μειωθεί το συστημικό κόστος της ενέργειας, να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, για τις ε, επιχειρήσεις αλλά και θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να απαλληφθούν η ρυθμιστική και μη ρυθμιστική φραγμή που αυτή τη στιγμή υφίστανται μεταξύ των ενεργειακών αγορών και να οικοδομηθεί η απαραίτητη υποδομή. Αυτό είναι απαραίτητο λοιπόν. Περαιτέρω όμως πρέπει οι εθνικές κυβερνήσεις να υλοποιούν, να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά τρόπο ορθό και ομοιόμορφο. Και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας ε, των αγορών ε, ενέργειας που να λειτουργεί σωστά υπό την επίβλεψη της Επιτροπής, θέματα που έχουμε συστήσει ήδη με τις υπηρεσίες ενέργειας, χωρίς το οποίο σύστημα δεν θα μπορούμε να έχουμε νέα ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και ιδιαίτερα νέες πρωτοβουλίες υπό τον τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τις εθνικές αρχές διάλογο σε σχέση με τις ευθύνες τους και κυρίως τα σημεία διασύνδεσης. Για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα. Θέλουμε ιδιαίτερα να δοθεί έμφαση στο σχέδιο, στους δύο, δύο αυτές για τις ε, αγορές μας. Η αποτελεσματικότητα, η μετάβαση περισσότερη βιωσιμότητα, μερικές φορές μπορεί να αντιμετωπίζονται ως προσκόμματα, ως βάρος για τις επιχειρήσεις είναι όμως όροι εκ των όνου κάνευ. Και όταν υπάρχει σαφής νομοθεσία με στόχους ξεκάθαρους μπορεί να δώσει τα κατάλληλα μηνύματα στις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα εξοικονόμηση πόρων. Αυτό μας λένε όλες οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνομιλούμε ότι θέλουν να έχουν ένα σαφές πλαίσιο που θα τους επιτρέπει και να προχωρήσουν και να επενδύσουν και να καινοτομούν ταυτόχρονα. Ε, πρόεδρε, βεβαίω περιμένω την καλή συνεργασία με του συναδέλφου. Είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να βρούμε καλέ συμβαστικέ λύσει και ότι έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συμβάλλει τα μάλα στην επίτευξη τη Ενεργειακή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρε, κυρίω που κρατήσατε το χρόνο, τήρησατε το χρόνο σα. Ο κύριο Τόμα εκ μέρου των Πρασίνων. Ο κύριο Τούρμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν περάσω όμως στην ουσία, θέλω να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που βλέπω να προτείνουμε τι μπορούμε να πράξουμε εδώ. Γιατί Κλείσαμε την έκθεση Χασάουτεκας με την, ε, για την ψηφοφορία με τις 900 τροπολογίες της. Πολύ εκτενής έκθεση. Είναι θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει τους τρεις μήνες, αποτελεσματικότητα στην προμήθεια κτλ. Τώρα τι θα κάνουμε θα περάσουμε σε μια σαββατικά παριθμών 2, θα πρέπει νομίζω και προτείνω να συμφωνήσουμε στους τομείς εκείνους, οποίους έχουμε ήδη συμβαστεί στην προηγούμενη έκθεση και να βρούμε τα σημεία τρυφής με το Συμβούλιο και την Κομισιόν γιατί διαφορετικά, εάν δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό να προτείνουμε στη συζήτηση αυτή, θα μα αγνοήσουν. Ο κύριο Πάτερσον ανέφερε πρώτο, Πέτερσεν, ανέφερε πρώτο την έννοια τη διακυβέρνηση. Τι είδου διακυβέρνηση, governance. Εμεί λέμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε περισσότερο εξευρωπαϊσμένο σύστημα, γιατί είναι πιο ε, μεγάλε οι οικονομίε κλίμακο, η σχέση κόστου αποτελέσματο. Άρα λοιπόν πρέπει να περιλάβουμε ένα κεφάλαιο στην έκθεση του ΙΟ, οποίο θα περιγράφουμε την υλοποίηση του συστήματος διακυβέρνησης και σε αυτό το σύστημα διακυβέρνησης πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει λόγο. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο, ο ρόλος του καταναλωτή, του, πολίτη, των πόλεων. Δεν γιατί ό,τι είδους νομοθεσία και να εισαγάγουμε, την καλύτερη δυνατή, το σύστημα αυτό πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη την κινητικότητά του, τις, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Εάν ας πούμε ένα μεγάλο αστικό κέντρο δεν μπορέσει να κινηθεί προς την έννοια της ε, εξοικονόμησης αποτελεσματικής χρήσης ε, του σωστού μείγματος, δεν κάνουμε τίποτα. Εξορθολογισμός λοιπόν μέσα στο σύστημα και ε, σχέση ενεργειακής ένωσης με τον πολίτη. Και κάτι ακόμη που ανέφερε και ο κύριος Γκιούρκη. Ποιος ηγείται των επιλογών των ενεργειακών στον κόσμο, η Ευρώπη. Εμείς έχουμε παθητικής ενέργειας ε, σπίτια, παθητική κινητικότητα, ανανεώσιμα. Πρώτοι εμείς. Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει όλα αυτά, αλλά τώρα κερδίζει έδαφος η Κίνα, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείες ο στρατός επενδύει τεράστια ποσά σε νέες τεχνολογίες. Πρέπει λοιπόν εμείς να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε την πρώτα καθεδρία μας. Ας κοιτάξουμε λοιπόν από τις ε, συμβαστικές λύσεις άδεγας πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε την ενέργεια, ε, μάλλον το πολίτη στο επίκεντρο των μελημάτων για την ενέργεια, την ε, πρώτο καθεδρία μας τεχνολογία, την διακυβέρνηση και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση όπως άλλωστε έχουν προσπαθήσει και ο κύριος Άδωρκας με όλους τους κοιόδης μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριο Σιλικιώτη της Σκουέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόπατσι για τη δουλειά που έχει κάνει. Ε, συμφωνώ με τον Κλούτ ότι μοιραία κάποια αρκετά ζητήματα θα τα επαναλάβουμε γιατί ήταν στην έκθεση Σοντάρκας ε, την οποία ε, πρόσφατα έχουμε εγκρίνει. Κατά την άποψή μας υπάρχουν σημαντικές παραλήψεις και έχουμε και διαφορές ε, σε όσα κατατίθενται σε αυτό το προσχέδιο. Ε, περιμένουμε να υπάρξουν τόσο συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να καταπολεμηθεί το νέο φαινόμενο της ενεργειακής στόχιας ε, και να δούμε ότι η ενέργεια είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση. Το δεύτερο είναι πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζονται ε, διασυνδέσεις και δημόσιες υποδομές ε, προς όφελες της κοινωνίας. Με τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενέργεια πρέπει να υπάρχει ενισχυμένος κρατικός έλεγχος ε, στις υποδομές και να προωθηθούν διεθνείς συνεργασίες στη βάση των όφελους. Το τρίτο είναι η ανάγκη να γίνει αναφορά για αξιοποίηση αποθεμάτων φυσικού αερίου που υπάρχουν σε κράτη-μέλη όπω στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Βεβαίω, χαιρετίζομαι την πρόταση που υπάρχει στο κείμενο για αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργεια. Ε, ωστόσο, διαφωνούμε με την πρόταση για αξιοποίηση όλων των ειδών ενέργεια που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, γιατί, όπω παραδείγματο χάρη τη πυρηνική ενέργεια, που ενέχει τεράστιου κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εμεί αντίθετα αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα ώστε να τερματιστεί η ανέργεια πυρηνικών σταθμών και ιδιαίτερα η ανέργεια πυρηνικών σταθμών σε ιδιαίτερα επικίνδυνε περιοχέ. Ε, έχουμε το παράδειγμα ε, της που γίνεται στην Τουρκία για την ανάγκηση του ΑΚΙΟΥ ενό ε, ε, πυρηνικού σταθμού σε σεισμογενή περιοχή, η οποία θα επηρεάσει γειτονικά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ιδιαίτερα προβληματική για μα στην έκθεση είναι η αναφορά στην ανάγκη τα κράτη-μέλη να έχουν μια φωνή στα ενεργειακά θέματα, καθώ και η έκκληση προ την Κομισιό να εξετάσει το πώ μπορεί να περιοριστούν οι εθνικές πολιτικέ. Οι εν λόγω προτάσει κατά ανάποψή μα καταστρατηγούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών και περιορίζουν τον κρατικό έλεγχο για τη διασφάλιση των συμφερόντων τη κοινωνία. Επίση, είμαστε, είμαστε αντίθετοι, αυτό βεβαίω υπάρχει και στην πρόταση τη Επιτροπή, για ενίσχυση του ρόλου τη Κομισιό στι Διακρατικέ Συμφωνίε μέσω τη συμμετοχή στι διαπραγματεύσει με τη διεξαγωγή αξιολογήσεων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, καθώ και με την κατάρτιση ρητρών απαγόρευση εξαγωγών και περιορισμού. Αυτά τη στιγμή που υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία είναι απομονωμένα από τα μεγάλα ενεργειακά δικτύα, τη στιγμή που υπάρχουν κράτη-μέλη με σημαντικέ ελλείψει στην ενεργειακή τροφοδοσία, θεωρώ ότι αυτό δημιουργά περαιτέρα προβλήματα και περιορίζει την εθνική ευελιξία στη διαχείριση ε, των εισαγών και εξαγών στα θέματα ενέργεια. Ε, εμείς ως ε, ε, θα στηρίξουμε, ε, ε, δεν θα στηρίξουμε την πρόθεση μια ενεργειακή πολιτική η οποία ελέγχεται από την Κομισιόν και τα ισχυρά κράτη-μέλη τη Ένωση, που θα περιορίζει την εθνική ευελιξία στη διαμόρφωση πολυδιάστατων και αποδοτικών διεθνών ενεργειακών σχέσεων. Μετά όσα σημεία έχω αναφέρει, βεβαίω θα καταθέσουμε ε, τροπολογίε για την βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, colleague. And the next speaker will be colleague Tamburan on εκ μέρου του Ευχαριστώ. Διαβάσαμε με προσοχή την έκθεση και σε πάρα πολλά σημεία διαφωνούμε. Πριν από λίγες ημέρες ε, λάβαμε με μεγάλη έκπληξη την είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αποφάσισε το 2050 να καταλήψει τα ορυκτά καύσιμα και εμείς ε, στην Ευρώπη ε, που φαίνεται να έχουμε ρηκτά καύσιμα κάτω από κάτι πέτρες, κάτι πολύματα και ένα θεός ξέρει πού, ε, ε, αγνοούμε την πραγματικότητα και δεν ε, βλέπουμε ούτε την ενεργειακή ούτε την οικονομική πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη στι Ηνωμένε Πολιτείε όπου η φούσκα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και του σχιστολιθικού πετρελαίου, αυτό το φυσικό αέριο το μη συμβατικό που υποσχόταν ε, δεν με τι θαύματα, ε, κατά πάσα πιθανότητα είναι μια φούσκα και μια οικονομική απάτη. Θεωρούμε ότι είναι λογικό να αφήσουμε κάποιους πόρους στο υπέδαφος για να τους χρησιμοποιήσουμε όταν θα είναι φαίνεται πιο βολικό να τις πουλήσουμε στην αγορά και να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Θεωρούμε ότι είναι παράλογο να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για θέρμανση κτηρίων όταν θα μπορούσαμε να μειώσουμε την ε, ε, χρήση φυσικού αερίου με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ενεργειακής απόδοσης. Μπορούμε να αλλάξουμε τις εισαγωγές του φυσικού αερίου και να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση για τα αιωλικά πάρκα, για ε, όλες τις υποδομές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Θεωρούμε... Ε, ε, πολύ σημαντικό το θέμα του πετρελαίου και επανέρχομαι σε αυτό. Για να κάνουμε ενέργεια μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Το πετρέλαιο είναι μια πολύ σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλών άλλων προϊόντων καταναλωτικών της βιομηχανοποιημένης κοινωνίας. Επομένως, ε, καλό θα ήταν να κάνουμε πραγματικά ένα άλμα στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί μας το ζητούν και οι πολίτες και η ιστορία, να κάνουμε μια αλλαγή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να φτιάξουμε αυτή την ενεργειακή ένωση πρωτό, πρωτίστως όταν ταξιδεύουν τα ηλεκτρόνια και όχι όταν ταξιδεύει υλικό μέσα σε αγωγούς. Και επίσης θεωρούμε ότι το ποσοστό διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών που προτείνεται είναι πολύ χαμηλό. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διασύνδεση. Και το Global Energy Sharing Network είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι παγκόσμιο και να κυκλοφορήσει και εκτός Ευρώπης διότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να έχουμε παγκόσμια χρήση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να σταματήσουν οι διακοπές που υπάρχουν μεταξύ εποχιακών ε, αλλαγών. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα την Ισλανδία για να χρησιμοποιήσουμε νέους ε, αγωγούς και νέα καλώδια και διατλαντικά και προς τη Δύση αλλά και γιατί όχι και προς Ανατολές. Να χρησιμοποιήσουμε όλους τους γείτονές μας από τη Μεσόγειο αλλά γιατί όχι και τη Ρωσία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που τουλάχιστον κατά την άποψή μου είναι ανησυχητική. Ευχαριστούμε συνάδελφε για τα σχόλιά σας και να ακούσουμε τώρα την άποψη της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Έχουμε τον Ιβο Μπέλετ, ο οποίος είναι συντάκτης της νομοδότησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και για την φιλοξενία. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφου ότι ο πρόεδρος Μπούζικ με τον πρόεδρο Λαβία έχουν καταλήξει μια πολύ καλή συμφωνία για τη συνεργασία των επιτροπών μας. Πρόκειται για εφαρμογή του άρθρου 54 του κανονισμού σε θέματα που είναι, κοινής, που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ε, των δύο επιτροπών, αλλά και μικτής αρμοδιότητας, ε, όπως σε παραδείγμα η απανθρακοποίηση ε, των μεταφορών και άλλα σχετικά θέματα. Να έχουμε λοιπόν καλή συνεργασία και στο μέλλον, ελπίζω. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια κύρια στοιχεία της έκθεσή σας πριν αναφερθώ στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφάλλοντος για την Ενεργειακή Ένωση. Λοιπόν, εμείς ε, έχουμε κοινούς στόχους μαζί σας, ε, όπως λέτε και στην έκθεσή σας, ε, ενεργειακή ασφάλεια, οικονομικές τιμές, ασφάλειες προμήθειες, ανταγωνιστικότητα για την βιομηχανία μας. Επίσης παραπέμπουμε στην γνωμοδότησή μας στο πλαίσιο 2030 Λέμε δηλαδή ότι μέχρι το 2030 θέλουμε να μειωθούν κατά 40% οι εκπομπές διοξιδίου του θερμοκηπίου. Κοινό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό όμως και να υπογραμμίζουμε και να υπενθυμίζουμε ότι προχωρούμε προς μια πολύ σημαντική διάσκεψη για το περιβάλλον στο Παρίσι στο τέλο του έτους. Ιδιαίτερο ρόλο αναγνωρίζουμε στο σύστημα ανταλλαγών εκπομπών ξέρουμε ότι προχωράμε σε μεταρρύθμιση του, ότι έχουμε φτάσει σε συμβαστικέ λύσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν από την Ολομέλεια για το απόθεμα σταθερότητας τη αγοράς, αλλά πολύ πιο σημαντικές αλλαγές θα προχωρήσουν σιγά σιγά για το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών. Περιμένουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις θερινές διακοπέ και πιστεύω ότι αυτά όλα θα είναι ε, καθοριστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση του λεφθέντος η απώλεια πηγών άνθρακα, ε, η διαρροή καλύτερα πηγών άνθρακα θα έχει τεράστιο κόστος για τη βιομηχανία. Στους τομείς εκτός του συστήματος ανταλλαγών επίσης θέλω να σταθώ. Πρόκειται για πολύ σημαντικό κομμάτι της, ε, Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, στο χώρο ο κατασκευαστικός και άλλοι, που όπως υπόθηκε πρέπει να ε, διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ήταν και στην προηγούμενη έκθεση Σάδοκα, τώρα θα έχουμε και σε αυτήν πιστεύω κάποια αναφορά ή θα πρέπει τουλάχιστον. Και ένα τελευταίο στοιχείο, η διασύνδεση με τι επενδύσεις του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ε, που φαντάζομαι ότι θα διατυπωθεί σε διάφορες τροπολογίες και επίσης θα ήθελα να επενθυμίσω την έκθεση Κούνα στην Επιτροπή των Μεταφορών ότι οι κανόνες για τις ε, ενέργειε μεταφορές και τις θαλάσσιες πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο παγκόσμιο προκειμένου να διφυλαχθεί και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανία Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Τώρα θα περάσουμε στου συναδέλφου με ένα μόνο λεπτό. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έχουμε 13 εγγεγραμμένους στον κατάλογο. Και ξέρετε ότι στι 10 πρέπει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Κύριο Μάνικα. Ďakujem, pán predseda. Ε, myslím si, že správa je veľmi dobrým východiskom a to, čo doplnili kolegovia... Je πολύ καλή η έκθεση, πιστεύω. Πολύ καλή σημείο κίνησης. Τα δε σχόλια που ακούσαμε σε σχέση με το κείμενο αυτό εδώ ε, νομίζω ότι δείχνουν πως προχωρούμε προς ένα καλό αποτέλεσμα. Η θέρμανση και η ψήξη είναι οι ε, ενεργειοβόρες χρήσεις. 40% της ενέργειας μας πάει στα ακίνητα και ως Υπουργό Ενέργειας Σλοβακίας στην προηγούμενη μου φοιτεία είχα υποστηρίξει ιδιαίτερα εξελίξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής μόνωσης των δημοσίων, δημοσίας χρήσεως κτηρίων μας, όπως τα σχολεία. Με αυτό θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε έως και 50 με 60% σε ενέργεια. Αν αυτό μπορούσαμε να το επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά τη ζήτηση σε ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια επένδυση καλή, δεν θα κοστίσει ιδιαίτερα γιατί έχει ε, επιχειρηματικό ή καλύτερα εμπορικό όφελος και οι απαιτήσει ενέργεια θα μειωθούν σημαντικά μαζί με την εξάρτησή μας από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω ιδιαίτερα την έκθεση του συναδέλφου Κρόβατσεκ. Ενέργεια λοιπόν και βιομηχανία. Με προβληματίζει λίγο το γεγονό, με εντυπωσιάζει λίγο το γεγονό ότι έχει γνωμοδότηση η Επιτροπή Περιβάλλοντο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η γνωμοδότηση είναι διεξοδική επικεντρώνεται σε διάφορα κέρια σημεία. Βλέπω προτεραιότητες ως προς τον χρήστη, τον πελάτη, αλλά και ως προς την κοινωνία γενικότερα και τη βιομηχανική χρήση. Αλλά εδώ βλέπουμε αλληλοαποκλειόμενες προτεραιότητες και γι' αυτό πιστεύω πρέπει να βρούμε μία λεπτή ισορροπία ένα συμβιβασμό θα έλεγα. Ο κύριος Μάνκα έφυξε το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας στη χρήση της ενέργειας. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όταν κοιτάμε το ΑΕΠ κατά κεφαλή, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Και υπάρχουν κράτη που έχουν θετικό ισοζύγιο και άλλα που έχουν αρνητικό. Ο πρόεδρος διακόπτει. Όχι, όχι πρόεδρε, μια τελευταία παρατήρηση ακόμα. Πρέπει το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών, το ETS, να γίνει πιο ορθολογικό στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζαρίνιο. <laughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κυρίως ε, για τη δουλειά του, αλλά θα ήθελα να πω ότι το αποτέλεσμα αυτή της αρχικής εκδοχής της έκθεσής του με ανησυχεί λίγο. Η Ενεργειακή Ένωση είναι ουσιαστική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει στρατηγικές και σαφείς επιλογές. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποδειγματική, καθορίζει ε, συγκεκριμένους πυλώνες βάσει επιστημονικών ενδείξεων. Οι πυλώνες αυτοί είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, η ενεργειακή απόδοση, ε, εφαρμοσμένες μέθοδοι. Η πρόταση κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και δεν είναι τόσο σαφής όπως ήταν η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει σημείο εστίασης και αποδυναμώνεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ίδια η, Ένωση, η Ενεργειακή Ένωση... έχει προβλήματα και μάλιστα αντιβαίνει στην αρχή της ε, πράσινης ανταγωνιστικής αγοράς η οποία θα μας οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας. Ελπίζω ότι με το έργο της Επιτροπής μας θα καταφέρουμε να ξαναβρούμε το σωστό δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Λεβαντόφσκι, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στο λεξιλόγιο. Το θέμα είναι να υλοποιηθεί κιόλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως αφορά και την ασφάλεια και τις ανταγωνιστικές τιμές γιατί εδώ πέρα είναι το μειονέκτημα της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση γιατί δεν έχει μόνο τα σημεία στα οποία συμφωνούμε αλλά προσπαθεί να κάνει και κάποια βήματα προόδου στην εξωτερική διάσταση. Εδώ πέρα ακριβώς είναι η ε, διαφορά γιατί υπάρχει ένας έλεγχος εξ αντε συμμόρφωσης. Και ακριβώς ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων ε, οπωσδήποτε κοστίζει περισσότερο από το να γίνεται ένας έλεγχος εκ των υστέρων. Αυτά σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Και πολύ καλές ε, παρατηρήσεις επίσης ε, ο κύριος Τοσανοφσκή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ενεργειακή Ένωση όπως όλοι ξέρουμε είναι κάτι το δύσκολο που μας περιμένει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των διαφορετικών συμφερόντων και της ε, διαφορετικής ιστορίας που υπάρχει. Ο κύριος ε, Κρυπάτσκι ε, συνέταξε ένα πάρα πολύ καλό κείμενο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί η χρήση των ερχόριων πόρων για να μειωθεί η εξάρτηση από ξένες πηγές. Δεν πρέπει επίσης ε, να απομονώνουμε κανένα κομμάτι ε, του ενεργειακού τομέα και θα πρέπει βέβαια να εκμεταλλευτούμε την έρευνα και την καινοτομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο κύριος Κάριντς. Ε, πρώτα απ' όλα στην προσπάθειά μας για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ξεχάσαμε λίγο την ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, είναι γεγονός πως το κόστος της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ που είναι και μεγάλος ανταγωνιστής. Ένας λόγος ε, για τον οποίο ε, είναι τόσο μεγάλο το κόστος είναι το ότι δεν έχουμε μια συνολική εικόνα. Παραδείγματο χάρη η Γερμανία πριν από λίγα χρόνια ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας παρά το ότι σαφώς δεν είναι η πιο ηλιόλουστη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα για να δούμε το θέμα του κόστους ε, στον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ, η κυρία Καλάς. Ευχαριστώ. Να πω βεβαίω πω εάν δεν ήταν ο, στο... ο τίτλος της έκθεσης δύσκολα θα καταλαβαίναμε ποιος ήταν ο στόχο γιατί εστιάζει πάρα πολύ στα κράτη-μέλη και τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και μια εσωτερική αγορά η οποία να λειτουργεί. Γιατί δεν κοιτάμε το ευρωπαϊκό συμφέρον. Η έκθεση δεν μιλάει αρκετά για την ανάγκη να υπάρξουν διασυνδέσεις και το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος ε, της ε, Κομισιόν. Και τέλος για τις ε, ενεργειακές για τις τιμές της ενέργειας. Εμείς έχουμε το παράδειγμα της Εστονίας που είναι ενταγμένη στην ε, σκανδιναβική ενεργειακή αγορά που μείωσε έτσι τις τιμές κατά 50%. Οπότε ένας ανταγωνισμός ο οποίος θα λειτουργεί μειώνει το κόστος. Οπότε εγώ θα ήθελα η έκθεση αυτή να εστιάσει περισσότερο στον ανταγωνισμό και στον στόχο της Ενεργειακής ε, Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γκρίφιν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση και θα διαμορφώσει το τοπίο για την επόμενη δεκαετία. Θα έχει επίσης αντίκτυπο στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, τις μεταφορές, την υγεία των παιδιών μας. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Δυστυχώς εδώ πέρα πάμε σε έναν ορίζοντα στον οποίο δεν είναι δεσμευτική η αποτελεσματική χρήση της ε, ενέργειας και δεν προωθείται η χρήση ανανεώσιμων πηγών. Αν είναι να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο θα βασίζεται σε, ε, και στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, της ΕΣΑ, τους πολίτες και της πόλης. Και τέλος πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και να κάνουμε κάτι για την ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και χρειάζεται να διευκρινιστούν, πιστεύω. Καταρχά. στην αρχή της έκθεση αναφέρεται ότι ο προσδιορισμό του μείγματο ενέργεια είναι αποκλειστική εθνική αρμοδιότητας. Μπορεί να έχει δίκιο ε, τυπικά ο εισηγητή, όμω τα ανανεώσιμα στην αποτελεσματικότητα και στην εσωτερική αγορά με βάση το 143 για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης λειτουργίας δηλαδή, ε, έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λοιπόν ε, άμεση σχέση η απόφαση, είναι ε, άμεσα επηρεαζόμενη η αγορά ενέργειας από τις αποφάσεις που θα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε. Και επίσης οι εγχώριες πηγές ενέργειας, οι οποίες άλλωστε αναφέρονται και ...την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να προσοριστούν πιο συγκεκριμένα. Ατομική ενέργεια θεωρείται και αυτή εγχώρια πηγή ενέργειας παρότι το 95% του ουρανίου προέρχεται από πηγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υδρορογμάτωση είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο καταγράφεται σε εγχώριες πηγές ενέργειας. Και θα ήθελα μια πιο σαφή τοποθέτηση εκ μέρους της Επιτροπής Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ρόιλ. Πρόεδρε, στη συζήτηση αυτή Φαίνεται να μας λέτε συνέχεια ότι πρέπει να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ της καλής και της κακής ενέργειας. Ε, όχι, εμένα με ενδιαφέρει να ακούω ποια είναι η πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και πώς μπορώ να είμαι πιο ανεξάρτητος ενεργειακά. Είναι όλο και πιο ακριβή, είναι πιο περίπλοκη, είναι όλο και πιο μεγάλη εξάρτησή μας από ενεργειακές πηγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω απαντήσεις λοιπόν και τα ερωτήματα δεν είναι καινούρια. Χρειαζόμαστε διαφοροποίηση στους τρόπους και στις οδούς μεταφοράς ενέργειας. Δεν χρειάζεται ε, στρεβλός ανταγωνισμός και τρίτον πρέπει οι δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη να διαδικτυωθούν περισσότερο. Γι' αυτό και η έννοια της δικτύωσης, η διαδικτύωση είναι το πιο καθοριστικό σημείο. Κάθε κρατος μέλος έχει τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματά του. Αν αυτά λοιπόν μπορούμε να τα συνδέσουμε έτσι ώστε να μειωθούν οι συνέπειες των μεν και να ενισχυθούν τα δε, τότε θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε συζητήσει ότι θα πρέπει να μειωθεί το κόστος με βάση την δικτύωση. Ωστόσο αυτό δεν εξασφαλίστηκε λόγω της ε, ε, ανεπάρκειας των επιλογών σε σχέση με τις ρυθμιστικές ε, διατάξεις και τελικά έχουμε λιγότερα. Ο κύριος Χριστοφόρου παρακαλώ. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σημερινό εισηγητή, τον κύριο αλλά και τον κύριο Σαουτάρκα για την προηγούμενη έκθεση για την εξαιρετική δουλειά που επέτυχαν όσον αφορά το ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, την οποία στηρίζουμε με όλε μα τι δυνάμει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να έχει ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία, πρέπει πρωτίστω να αξιοποιήσει τα δικά τη φυσικά αποθέματα, είτε είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε σε άλλε περιοχέ, στηρίζοντα αυτέ τι υποδομέ. Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, είναι αδιανόητο να επιτρέπεται ανέγερση σταθμών όπω το ΑΚΚΙΟΥ εκεί και όπου υπάρχουν σεισμογενεί περιοχέ. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο και πλήττει ακόμα και την πολιτική για την πυρηνική ενέργεια. Οπωσδήποτε πρέπει και εμεί να επικεντρωθούμε στα ζητήματα τη καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια και πρέπει να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο ω Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιδείξουμε την ευαισθησία μα. Τέταρτο, νομίζω ότι πρέπει η ΑΠΕ που ήταν, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να τον έχει και αν μπορεί ακόμα να αυξήσει και το στόχο από το 20% και να υπάρξει προ αυτήν την κατεύθυνση ανάπτυξη, επικέντρωση για την καινοτομία και την έρευνα. Και τέλο, ήθελα να πω ότι πρέπει επιτέλου να επικεντρωθούμε σημαντικά όχι μόνο σε εκθέσει αλλά και σε πράξει για τα θέματα τη ενεργειακή ασφάλεια και τη ενεργειακή αυτάρκεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Short remarks. Σας ευχαριστώ. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Βέλσντερφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Γκρομπάτση και την πάρα πολύ καλή έκθεση. Να τονίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα η ε, Ενεργειακή Ένωση είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο ζήτημα και αυτό που έχει σημασία, όπως είπαν κάποια κράτη-μέλη ε, είναι η εφαρμογή της. Θα αναφερθώ λοιπόν σε κάποια πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα η έκθεση Σάντεγκας. για την ε, σημασία της ε, ενεργειακή Ένωσης. Δεύτερον, για την ανταγωνιστικότητα και το κόστος ενέργειας, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κάναμε μία μελέτη πέρσι και θα κάνουμε άλλη μία. Και βεβαίω θα δούμε τις διαφορές μεταξύ των τιμών χοντρική και λιανικής και μεταξύ κρατών ε, μελών. Και είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τι τεράστιε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά ε, στην πλευρά της λιανικής ε, λόγω φόρων Όσον αφορά τώρα την ε, ασφάλεια παροχής, η Κομισιόν θα κοιτάξει το θέμα της στρατηγικής θέρμανσης και ψήξης αλλά και της αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και πριν από το καλοκαίρι θα φέρουμε ένα έγγραφο διαβούλευσης για να παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες για το πώς θα πρέπει να έχει αγορά. Τέλος, για την ε, διοίκηση, την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, συμφωνώ. Ε, προφανώς ε, βεβαίως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους εταιρείς μας για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Κύριε Σίγητα, στην αρχή είχατε 12 λεπτά, τώρα ένα λεπτάκι για τις παρατηρήσεις σας. Ε, δεν έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ε, πολλές τους παρατηρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να συνομιλούμε για να βρούμε κοινέ λύσεις. Και γι' αυτό πολύ πρόθυμα θα ακούσω κάθε νέα πρόταση. Σας καλώ στη συνεργασία λοιπόν. Σας καλώ στην αναζήτηση συμβιβασμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ενέργειας που είναι και το πιο σημαντικό θέμα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Σπουδαία, τα είπατε. Ευχαριστούμε για την έκθεση, ευχαριστούμε τους και ηγητές για τη συζήτηση. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 4 Ιουνίου και όχι 3. 4 Ιουνίου, έχετε μια μέρα παραπάνω του 2015, 12 το μεσημέρι. Θα πρέπει βεβαίω να ληφθεί υπόψη και η γνωμοδότηση Επιτροπή του Περιβάλλοντος. και την εβδομάδα που θα έχουμε τις ψηφοφορίες το Σεπτέμβριο θα ψηφιστεί για να εξεταστούν οι τροπολογίες στο μεταξύ 15-16 Ιουλίου. 4 Ιουνίου λοιπόν τροπολογίες. Στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση για την Ενεργειακή Ένωση. Είπε και ο εισηγητής ότι πρόκειται για το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ε, θητείας μας. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες με αρχικά δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν τα συστήματα δουλεύουν. Τοποθετήστε τις κάρτες σας παρακαλώ στις σχισμές. Δουλεύουν όλα. Και η ερώτηση που θέτω πάντα, σας αρέσει η Επιτροπή Ένβη. Όχι η Ήτρε, μην πείτε για την Ήτρε. Η ερώτηση λοιπόν στην οποία πρέπει να ψηφίσετε είναι, σας αρέσει η Άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. Είναι σημαντικό να μην το ξεχνάω. Ο Ιβο Μπέλετ είναι εδώ. Να του στείλετε ένα email παρακαλώ. Να έρθει αυθόρυ και παραχρήμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι συνάδελφοι. Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και νήσων Φαρόε. Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Ένας πλεονάζων από το σοσιαλιστές. Ένας υπεράριθμος. Ναι, ναι, πρώτη φορά στην ιστορία έχετε δίκιο. Εγκρίνεται. Δεύτερο θέμα, συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας Συνδίας, άρχεται ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από τους Σοσιαλιστές Πέρας, εγκρίνεται. Επόμενο θέμα, Συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τη Ομοσπονδία της Ελβετίας και την Ευρωπαϊκή Ατομική, ε, Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης προς μια κυκλική οικονομία. Ο Μπένεντεκ Γιάβορνο, εισηγητής, Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4α συμβαστική υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Η 4α συμβαστική τροπολογία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4β υπέρ. Κατά. Για άλλη φορά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. 4β συμβαστική. Πέρας. Εγκρίνεται και πάλι. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Συμβιβαστική 5. Πέρασε. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 45 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε παρακαλώ. Τη 45. Τροπολογία 45 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Προφορική τροπολογία του εισηγητού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η εξή η προφορική μας τροπολογία. Υπογραμμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση ε, θεμητού ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ε, απόβλεπα, απόβλητα ακόμα και αν πρόκειται για δημοτικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την αποκομιδή των αποβλήτων. Ε, παρακαλώ να δίνει υποστήριξη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Η συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά Εγκρίνεται, αλλά σε απολυθεύσουμε τη συμβαστική 10. Πέρας. Εγκρίνεται. 57 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας επαληθεύσουμε. 57. Πέρας. Υπεράριθμος 1 στο, στους σοσιαλιστές. Πέρας. Απερίφθη. Απερίφθη. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Την 93. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 16 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε την 105 ηλεκτρονικά πέρας απερίφθη συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο άρχεται ψήφισαν όλοι Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριο Μπέναντεκ Γιάβου. Αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτό ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία μας και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, αμέσως νομίζω. Ναι, ναι, μπορούμε, μπορούμε. Πάνω στην ώρα ήρθατε. Αγαπητοί φίλοι, αν θέλει κάποιος να αποχωρήσει, λυπάμαι βέβαια που φεύγετε, αλλά σας παρακαλώ ησύχως, χωρίς πηγαδάκια. Δεν με ακούει και κανείς. Uh, Ευχαριστώ, συναδελφοί, κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ πολύ να σταματήσουν τα πηγαδάκια. Συνάδελφοι εδώ δεξιά. Ησυχία παρακαλώ. Λυπούμαστε που φεύγετε μεν, αλλά σας παρακαλώ πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε τις δυνατότητες της έρευνας και της καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία. Έχουμε την εξέταση των τροπολογιών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή είναι απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία και υπευλήθησαν 223 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Η Επιτροπή μας θα λάβει και γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Αλίας. Θα μας στείλουν λοιπόν τις γνωμοδοτήσεις τους. Συνολικά έχουμε περίπου 40 λεπτά προς Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο εισηγητής ε, ο, είναι ο κύριος Φερέιρα από την ΚΟΕ. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να μας κάνετε την αρχική σας παρέμβαση. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσους θα συνεισφέρουν στην βελτίωση αυτής της έκθεσης έχουν υποβληθεί περίπου 220 τροπολογίες, κάτι παραπάνω και νομίζω ότι ε, έχουμε τις προϋποθέσεις προκειμένου να εξετάσουμε τις διάφορες συμβαστικές προτάσεις. Καταρχάς, ε, στην πρώτη συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές φάνηκε σαφώς ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν συμβιβαστικές τροπολογίες και χωρίς να καθυστερήσω περαιτέρω θα ήθελα να επισημάνω κάποιες ε, από τις πιο σημαντικές ε, πτυχές. Ε, οι οποίες είχαν και τις περισσότερες τροπολογίες άλλωστε. Από ό,τι διαπιστώνω υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα επί του οποίου καλό θα ήταν να ακούσουμε και λίγα περισσότερα. η άποψη των, των συναδέλφων αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τη δημιουργία ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οργανισμός ο οποίος θα έχει διάφορες αρμοδιότητες όσον αφορά τη γαλάζια οικονομία. Δεν προτείνεται ακριβώ ε, κάτι συγκεκριμένο, αλλά ε, η ιδέα δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα ε, υπηρεσία. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και ε, μια υπηρεσία μέσα σε ένα προϋπάρχοντο οργανισμό για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες αρμοδιότητες και κάποια ε, ε, θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένα και βρίσκονται ε, στην αρμοδιότητα διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών. Θέλουμε να προωθήσουμε με κάποιο τρόπο τη γαλάζια οικονομία και ε, βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή των κρατών μελών και δέσμευση και των κρατών μελών και των αρχών τους. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα εκτός και αν πρόκειται για κάποιο πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν και ίσως ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη της ανάπτυξης των δυνατοτήτων ε, της γαλάζιας οικονομίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, επίσης και κάποιες τροπολογίες που αφορούν το θέμα της εκμετάλλευσης των παράκτιων ορυκτών πόρων Υπάρχουν και διεστάμενες απόψεις, οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση εδώ, διότι ερίζουν οι απόψεις, ε, έχουμε κάποιες τροπολογίες οι οποίες δεν θέλουν να καλύπτονται καν ε, με την, από την έννοια αυτή και κάποιοι άλλοι έχουν υποβάλει προπολογίε που θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι τομέα προτεραιότητα στη γαλάζια οικονομία το συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, υπάρχουν και κάποιες θέσει που θέλουν να συμπεριλάβουν μεν ε, τις δραστηριότητες αυτές ε, στη γαλάζια οικονομία αλλά ε, να μετριαστούν οι συνέπειές της με κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν την συντήρηση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επόμενο ζήτημα. Δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Γνωρίζουμε τις διάφορες ε, θέσεις επί του ζητήματος, πρόκειται για το περιβόητο CCS και ίσως θα έπρεπε να ακούσουμε λίγο και τις απόψεις των συναδέλφων επί του ζητήματος και κυρίως όσον αφορά τις τροπολογίες που κατέθεσαν για τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα. Στη συνέχεια έχουμε και διάσταση απόψεων όσον αφορά την εκμετάλλευση των πόρων ε, στη γαλάζια οικονομία. Αφενός ε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, πιστεύουν ότι κατά προτεραιότητα θα πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια άλλη προσέγγιση προτείνει να σεβαστούμε την ε, ποικιλομορφία των προτεραιοτήτων ε, και των διαφόρων επιλογών μεταξύ των κρατών μελών. Ε, προφανώς και μεταξύ των κρατών μελών θα είναι διαφορετική ε, σε κάθε θέμα, όχι γιατί είναι διαφορετική απαραίτητο ή πόρη, αλλά οι προτεραιότητες μπορεί να διαφέρουν από κράτο μέλο σε κράτο μέλος. Μπορεί να είναι διαφορετική ε, η προσέγγιση του κάθε κράτο μέλο, οι πρώτε ύλε που διαθέτουν και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και ότι υπάρχουν τελείω διαφορετικέ περιπτώσει, επομένω, προτείνονται και τελείω διαφορετικέ επιλογέ και ίσω αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στους κοιόδης εισηγητές. Η κυρία Σπυράκη, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Υπήρξαν πολλές ε, τροπολογίες ε, οι οποίες κάλυπταν το ίδιο ζήτημα και ίσως ε, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να βρούμε κάποιο κοινό έδαφος σε κάποιες. Έγινε μια συνεδρία των σχεδόν εισηγητών ε, στις αρχές της εβδομάδος, όπου καθορίσαμε τα βασικά θέματα επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Καταρχάς, το θέμα της δημιουργίας ενός νέου οργανισμού. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πρόταση, όπως γνωρίζετε, η θέση του ΕΛΚ είναι συγκεκριμένη. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ένας υπάρχον οργανισμός να αναλάβει τα θέματα της έρευνας και θαλασσίων δραστηριοτήτων και κάποιες άλλες ε, οργανισμούς θα μπορούσαμε να τους συγκεντρώσουμε αν βελτιώσουμε, μπορούμε να βελτιώσουμε το τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Αυτή είναι η θέση μας, ε, αυτό άλλωστε προκύπτει και από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε την ε, υπάρχουσα χρηματοδότηση υπό μία σκέπη. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία προτείνονται στον ορίζοντα 2020 που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καινοτομία και τη γαλάζια οικονομία. Θεωρούμε επίσης ότι όσον αφορά τη χρηματοδότηση θα πρέπει ε, κυρίως να σχεδιάσουμε τη χρηματοδότηση τομέων γαλάζιας ανάπτυξης. Ε, θεωρούμε ότι αν επικεντρωθούμε σε κάποιες στοχευμένες προτεραιότητες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνέπειες της χρηματοδότησης, ιδίως αν είναι χαλεπή η πόρη μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική για όλες τις περιπτώσεις και να επιβάλλουμε συγκεκριμένε προτεραιότητες στα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι κάθε κράτος μέλος να καθορίσει σαφές τους στόχους και τις προτεραιότητές του, ώστε να βελτιωθούν οι συνέπειες της χρηματοδότησης που θα λάβει. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η γαλάζια οικονομία είναι μόνο μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το παρόν. Δεν είναι στρατηγική. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει στρατηγική. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους και το προσωπικό για τις συμβαστικές τροπολογίες και όσον αφορά τα πιο πιεστικά ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιο κοινό έδαφο. Και ένα σύντομο σχόλιο για τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Όπως ξέρετε, το ΕΛΚ είναι κατά της περαιτέρω χρηματοδότηση επί του ζητήματος. Ευχαριστώ. Thank you very much. And on behalf of... Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους σοσιαλδημοκράτες, η κυρία Μίριαμ Τέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει και για την πρώτη συζήτηση που κάναμε για το σε ποια ζητήματα μπορούμε να συμφωνήσουμε και το ε, σε ποια ζητήματα μπορούμε να έχουμε ένα κοινό μέτωπο αλλά μπορώ να πω πως μπροστά μας έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την γαλάζια οικονομία σε ολόκληρη την Ένωση. Εγώ θεωρώ πως για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη της της οικονομίας χρειάζεται μια συνεκτική θαλάσσια και ναυτική δράση. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ λίγο πιο λεπτομερώς στην πρότασή μας για μια σχετική υπηρεσία, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και τα ξέρει αυτά και συζητής. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε ακόμα μια υπηρεσία, αλλά το πώς θα μπορέσουν όλες οι σχετικές υπηρεσίες και διευθύνσεις να στεγαστούν κατά από μια κοινή στέγη. Θεωρώ πως χρειάζεται μια συνεκτική τέτοια στρατηγική που θα διατηρούνται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και θα υπάρχει συντονισμός. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν ξέρει η δεξιά τύπη ή η αριστερά μας όσον αφορά την κιανή οικονομία και νομίζω πως είναι αυτό κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ε, θα κανονίσουμε το πού θα είναι η έδρα, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε από τις αρχές ότι πρέπει να είναι κάτω από μία στέγη όλες οι σχετικές υπηρεσίες και νομίζω πως αυτό μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Αναφέρουμε επίσης τη χρηματοδότηση. Θεωρούμε πως και η Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν ε, επαρκή χρηματοδότηση για να υπάρχει συνέχεια και προβλεψιμότητα, αλλά για εμάς είναι απολύτως απαραίτητο να μην ε, διακινδυνεύσουμε αυτή τη στιγμή την συνέχεια των υφιστάμενων προγραμμάτων αλλά και να μην υπάρχει σπατάλη πόρων και καταργησή έργων γιατί σε τελική ανάλυση θα καταλήξουμε εκεί ακριβώς. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που θα ήθελα να τονίσω ικανοποιήθηκα για το ότι συμφωνούμε για το ότι δεν ε, υπάρχει μία ενιαία λύση γιατί μιλάμε για θάλασσες και ωκεανούς με μεγάλη ποικιλομορφία και τέλος πρέπει να αναφερθεί η έλλειψη πληροφοριών για τους ωκεανούς, για τους πόρους και την αλληλεπίδραση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ κύριος Γκρομπάρτσικ για το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος είναι γνωστός για το πως συνεισφέρει στα θέματα αυτά. για τα ζητήματα αλληλείας, συμπροστασία προστασία των μικρών ληφτικών κοινοτήτων και βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρει για την σχετική στρατηγική. Πρώτα απ' όλα αναφέρει την έλλειψη κοινής πολιτικής ε, θαλάσσιας διαχείρισης. πρέπει νομίζω να αποκαταστήσουμε την, τον κλάδο των ναυπηγείων. Ένα άλλο θέμα βέβαιο είναι οι θαλασσίες μεταφορές. Ε, ένα στόχο ο οποίο δεν έχει βρει μέχρι στιγμή σε σωστή εφαρμογή. Κατόπιν είναι η εξερεύνηση των θαλασσών. Υπάρχει λοιπόν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, κάποιες λύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές και θα μας δώσουν την ε, δυνατότητα να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι στις ε, προμήθειές μας. Και αυτό θα επηρεάσει και την πολιτική του κλίματος και ευχαριστώ τον Τζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ταμπουράνο για το EFDT. Το σχέδιο έκθεση του εισηγητή αποτελεί καλό εφαλτήριο. Συμφωνούμε με την ε, άποψη ότι ε, η χρηστή χρήση των θαλάσσιων πόρων δεν ε, συνάδει με τη χρήση του οικοσυστήματος. Θα πρέπει πρωτίστως να κοιτάμε την προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Τη μάχη και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές δηλαδή. Για αυτές τις αρχές όμως πήγαμε πέραν των παρατηρήσεων του συναδέλφου στις τροπολογίες μας, διότι θεωρούμε ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την περιγραφή και την εκμετάλλευση των ε, ορυκτών πόρων που έχουν ε, ε, σύντομη διάρκεια, δεν δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα και λοχεύει ο κίνδυνος να καταστρέψουν ε, τον βήθο της θάλασσας που σημαίνει ότι αυτό θα είναι εις βάρος για τις μελλοντικές γενναίες. Ζητάμε λοιπόν μορατόριουμ για όλες τις διαδικασίες εξόριξης μακροπρόθεσμα. Επίσης θεωρούμε ότι η εκμετάλλευση της γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να βαίζεται σε βιώσιμες οικονομίες πολιτικές που θα πρέπει να διαφυλάξουν και την μελλοντική γενεά αλλά και την παρούσα και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βασιστούμε στα οικοσυστήματα βάσει του άρθρου 190 της Συνθήκης της Λισαβόνας και της ε, ε Συμφωνίας του Ριό. Και ελπίζω να υπάρξουν σημεία σύγκλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχει ιδιαίτερη σημασία πιστεύω εμάς, για μας το θέμα αυτό. Και μια καλύτερα τα δύο τρίτα της Φιλίου από νερό, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι είδους τεχνολογία χρειαζόμαστε και για την εκμετάλλευση των βυθών. Είναι κάτι το οποίο έχει εντάξει ως μελέτη η Επιτροπή των Οικονομικών ε, στο σχεδιασμό της το deep sea exploitation δηλαδή, την εκμετάλλευση των θαλασσιών βυθών, ώστε να ξέρουμε τι είδους επιλογές υπάρχουν και η νομοθεσία πώς μπορεί να τις αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό. Πιστεύω ότι θα πρέπει και ο εισηγητής και οι εισηγητές να κοιτάξουν τις μελέτες αυτές, να λάβουν υπόψη τις επιλογές που προσφέρουν, διότι είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να έχουμε υπόψη πάντα τα επιστημονικά στοιχεία. Uh, uh Σας ευχαριστώ. Έτερος. Όχι. Έχουμε μέρους Επιτροπής. Κύριος Μπέιτς. Η Γενική Διεύθυνση Μάρε των θαλασσών. ευχαριστώ πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, τους συναδέλφους, τη Γενική Διεύθυνση για την έρευνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια. Ιδιαίτερα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έγγραφο αυτό που αναφέρεται στην καινοτομία. Βεβαίως θα μελετήσουμε τα, ε, τους προβληματισμούς και τα, επιχειρήματα που εγέρθηκαν. Δεν έχουμε κατασταλάξει. Είμαστε σε σχέδιο ασμό ακόμη. Άρα δεν θα μπορέσω να επισελθώ σε λεπτομέρειες ε, για να πω το σημείο φι μας αρέσει, το σημείο χ δεν μας αρέσει. Έχουμε την ε, ανακοίνωση του 2014 που έχει σαν στόχο τον εστιασμό στην καινοτομία και την μπλε λεγόμενη οικονομία θέματα δράσεως ε, όπως ε, εγκαθίδρυση επιστημονικών ε, και επιχειρηματικών φόρουμ. Φέτο προβλέφθηκε ένα σχετικό φόρουμ στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή ημέρα της ναυτιλίας. Αντίστοιχες δράσεις έχουμε στο σχεδιασμό μας και προωθούμε θέματα που έχουν να κάνουν παραδείγματι με μια υπηρεσία που θα ασχολείται μόνο τα θέματα της μπλε οικονομίας. Είναι ενδιαφέροντα, μεν, αλλά δεν ε, υιοθετούμε την ίδια προσέγγιση. Στο σχέδιο με τις τροπολογίες βλέπουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ορυκτά από το θαλάσσιο βυθό. Είναι κάτι το οποίο θα μας επαναφέρει στην πρόταση του 2012 όπου είχαμε πει πως δεν θα πρέπει να ε, εκδιωχθούν ή να περιθωριοποιηθούν από τον τομέα της εκμετάλλευσης των θαλασσίων βυθών οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια πιλωτική δράση. Αυτή τη στιγμή μόνο κοιτάμε να αναλύσουμε, να αναλύσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξόριξη από τους θαλασσιούς βυθούς, ώστε να έχουμε υπόψη μας ε, τα, όλα τα στοιχεία τα σχετικά. Αποθήκευση άνθρακα δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων μας. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση για την έρευνα έχουν σχόλια. Είναι της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας. Πάντως γενικά είναι ένα θέμα το, για το οποίο έχει εκφραστεί υποστήριξη και στο παρελθόν και μάλλον, αν δεν με εγώ, ε, και στο παρόν. Επίσης ένας εκ των ομιλητών αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πολλές ήταν οι επικαλυπτόμενες τροπολογίες, όντως, μία από τις ε, προτινόμενες τροπολογίες ε, προτείνει κάτι το οποίο δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέλω να σας το επισημάνω. Έχει να κάνει με τη γεωργία, και συγκεκριμένα η τροπολογία 176, παράγραφος 16, που απευθύνει η έκκληση για την υποστήριξη στη μετάβαση από τις παραδοσιακές γεωργικές ή συμβατικές γεωργικές μεθόδους στην βιολογική, ε, παραδείγματι γεωργικά συστήματα κλειστής κυκλοφορίας. Εδώ στην ε, βιολογική υδατοκαλλιέργεια έχουμε μια απόφαση του 2006 που δεν το επιτρέπει να εισαχθούν τέτοιες λύσεις γιατί ήταν ένα σύστημα το οποίο προσέγγισε πάρα πολύ το σύστημα της ε, εκμετάλλευσης. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα ε, ίσως υπάρχει περιθώριο να ξανανοίξει και να συζητηθεί. Πάντως όπως ισχύει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν επιτρέπει αυτή την προσέγγιση για τη βιολογική παραγωγή. Με τα σχόλια αυτά νομίζω μπορώ να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν ξαναδώσω τον λόγο στον εισηγητή να σας ενημερώσω πως σε 15 λεπτά θα έρθει εδώ ο κύριος Έτιγκερ σε 10-15 λεπτά και όπως βλέπετε η αίθουσα είναι άδεια. Και ήταν παρόλα αυτά στην ημερήσια διάταξη η επίσκεψη Έτιγκερ. Με πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ο δικός χάρτης ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακή αγοράς. Πολύ σημαντική συζήτηση. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να τηλεφωνήσετε τους αδέλφους να έρθουν. να έρθουν σε 10-15 λεπτά που θα ξεκινήσουμε. Πάρτε σε ένα τηλέφωνο γιατί η εικόνα είναι κάπως απογοητευτική. Ο κ. Ισοπέτροπος λοιπόν θα είναι εδώ σε 10-15 λεπτά. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τον εισηγητή μας. 15 λεπτά λοιπόν έχετε τον λόγο για 15 λεπτά. Ίσως ο κύριος Γκομπάτζικ μπορεί να προσθέσει κάτι στην προηγούμενη έκθεση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, αν απαντούσα ε, θετικά ίσως να αδειάζει κι άλλο η αίθουσα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτές τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις και οπωσδήποτε θα καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις που θα αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Αυτά σχετίζονται και με αυτό το οποίο μόλις είπε η Κομισιόν. Υπάρχει νομίζω λοιπόν εδώ πέρα μια μεγάλη συνένεση. Ισχύει λοιπόν η διαπίστωση ότι η προσέγγιση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ περιοριστική. Η ανακοίνωση την οποία βγάλαμε ότι δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και εδώ πέρα έρευνα και ανάπτυξη είναι μια ανακοίνωση που επικεντρώνεται σε ένα πάρα πολύ μικρό τομέα εξορίξεις στη θάλασσα, βιοτεχνολογία και τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να επεκταθεί αυτό το θέμα με τρόπο πιο ολοκληρωμένο και για μία σειρά τομέων που ανήκουν επίσης στην γαλάζια οικονομία. Οι δε κλάδοι αυτοί προστίθενται στους παραδοσιακούς ναυπηγεία, ηχθειοκαλλιέργεια και τα που επίσης δεν πρέπει να τα ξεχνάμε σε για, για μια αναπτυξιακή στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, συνάδελφε για την εκθεσή σας. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα για μας, ε, η γαλάζια οικονομία. Ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης 16 Ιουνίου 2015. Έχουμε συνολικά 223 τροπολογίες. και νομίζω ότι σε τέσσερις εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ο χάρτης πορείας για την ολοκλήρωση της ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ε, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ ο κ. Ζέτιγκερ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, α αρχίσουμε. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο που ήρθε στην Επιτροπή μα. Όπω είχαμε συνηθίσει και στην προηγούμενη θητεία, είναι απόλυτα φυσιολογικό να έρχεται στην Επιτροπή Βιομηχανία ο Επίτροπο Έτιγκερ για να συζητήσουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά, αλλά βέβαια όλα αλληλένδετα είναι διαφορετικό γιατί μιλάμε για την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά προκειμένου να δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Ο δικός χάρτης λοιπόν για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Ανταλλαγή απόψεων. Με εσάς κύριε Επίτροπε. Υπεύθυνο για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο δικός χάρτης. Ο δικός χάρτης είναι και αυτός πολύ σημαντικός για μας, όχι μόνο ε, μια ιδέα γενική μια στρατηγική, αλλά ως στοιχείο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της ιστορικής ψηφιακής αγοράς και για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. προσδοκία μας είναι από εσά να ακούσουμε τα των δράσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως όσον αφορά ίσως τους πυλώνες υπαριθμών 2 και 3 της στρατηγικής σας. Διαλειτουργικότητες. Γιατί έχουμε τρεις κύριους πυλώνες, ξέρετε, με τη σειρά που τους καταγράφει η ανακοίνωση, ο πρώτος πυλώνας αφορά περισσότερο τις άλλες επιτροπές και κατά την ε, Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς περισσότερο από τις άλλες. Ο δεύτερος και ο τρίτος όμως πυλώνας είναι πυλώνες δικών μας αρμοδιοτήτων και ως εκ τούτου θέλουμε να ακούσουμε κάθε πληροφορία σχετική με, τον, με το φύλλο πορείας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής εσωτερική αγοράς. Έχετε τον λόγο κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπούζεκ, κύριε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξαναμιλήσουμε και αυτό το οποίο ανακοινώνουμε με το πακέτο της ε, Κομισιόν θα είναι μια σειρά κοινών δράσεων που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πηγαίνουμε προς έναν δρόμο ε, εξορθαϊσμού της ε, ψηφιακής πολιτικής για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και χρειαζόμαστε θα έλεγα μια διαφορετική κουλτούρα και ταχύτητα εργασίας στον ψηφιακό τομέα. Κανένας άλλος τομέας δεν αλλάζει τόσο γρήγορα. Με τεχνολογίες που εξελίσσονται ραγδαία. Γι' αυτό πέρα από το περιεχόμενο θα πρέπει να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα. Είμαστε πάρα πολύ αργοί. Η κουλτούρα μας, πράσινο βίβλος, ε, απαντήσεις, ε, λευκή βίβλος, ε, ανακοίνωση, νομοθεσία και επαναδιατύπωση και μετά μπλοκάρει ένα χρόνο το θέμα στο κοινοβούλιο και δεν υπάρχει στο Συμβούλιο μου συγχωρείτε και να υπάρχει εντολή και μετά πάμε σε τριμερή διάλογο και αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα όσον αφορά το πακέτο αυτό. Μέχρι να φτάσει να εφαρμοστεί κάτι στο, στον πραγματικό κόσμο περνάνε 7 χρόνια. Και δεν θα περιμένει κανείς 7 χρόνια. Οι άνθρωποι θα κάνουν την δουλειά τους και απλά εμείς γινόμαστε γελοί και να με συγχωρείτε. Τι να σας πω, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά, ούτε στην ε, γεωργία, ούτε στην ε, κτηνοτροφία, ούτε στην κλιματική πολιτική. Είναι τραγικά αργή αυτή η φρόνη αντίδραση και οι Ευρωπαίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν το τρένο αυτό της ε, ψηφιακής επανάστασης και να μείνουν πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε πιο γρήγορα, να ερευνούμε ε, και να κινούμαστε γρηγορότερα και να επενδύουμε γρηγορότερα στις υποδομές και να παράγουμε και γρηγορότερα νομοθεσία. Αυτό θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ως βασική πρόκληση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά δημοκρατικά όργανα. Ποια είναι λοιπόν τα σημεία, τα κύρια για την στρατηγική μας για τον εξευρωπαϊσμό της ψηφιακής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα μια εσωτερική ψηφιακή αγορά. Γιατί, γιατί πρώτον η Ευρώπη πέραν από μία κοινωνία αξιών και μία κοινότητα ε, οικονομική ήταν πάντα μία εσωτερική αγορά υπηρεσιών ε, και αγαθών Ισχύει αυτό για αγαθά και για ψηφιακές υπηρεσίες, για αυτοκίνητα και για ψηφιακά προϊόντα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχει πάρα πολύ... είναι απολύτως αναγκαία η εσωτερική ψηφιακή αγορά. Αν φτιάχνει κανείς αυτοκίνητα έχει τεράστιο κόστο ανάπτυξης και κόστος παραγωγής. Όταν φτιάχνει κανείς τρόφιμα έχει άδεια, έχει κόστος άδεια, ε, κάποιο κόστος ανάπτυξης στην αρχή και παραγωγής. Αλλά οι εφαρμογές ε, έχουν υψηλό κόστος ανάπτυξης, αλλά όταν είναι έτοιμη η ψηφιακή υπηρεσία, το ε, ερώτημα το αν έχει κανείς 100 πελάτες ή ένα εκατομμύριο πελάτες είναι μετά διάφορο. Το οριακό κόστος είναι σχεδόν μηδέν. Και ακριβώ εδώ πέρα αυτό συνδέεται, παραδείγματο χάρη, ε, και είναι ανάλογο με αυτό το οποίο γίνεται με την ηλιακή ενέργεια. Δηλαδή είναι μεγάλο το αρχικό κόστος ανάπτυξη, αλλά αυτή τη στιγμή μπει το πάνελ στην οροφή, το κόστος παραγωγής ε, είναι σχεδόν μηδενικό. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε ένα μέγεθος αγοράς, γιατί αυτοί οι οποίοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα είναι 28 ε, κατακαιρματισμένες αγορές θα είναι τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου που είναι μεγαλύτερη από τη ΣΥΠΑ. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στα μάτια ε, και να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε ΙΠΑ, Κορέα, ε, Ιαπωνία και Κίνα. Κάθε αγορά επίσης χρειάζεται κάποιες δυνατότητες μεταφοράς. Εδώ πέρα δηλαδή αυτό ισχύει, μιλάμε για ταχύτητα, ποιότητα και δυνατότητες. Είτε μιλάμε για δρόμους, ε, αεροδιαδρόμους, ε, είτε για θαλάσσιες οδούς και το ίδιο ισχύει και για τις ψηφιακές οδούς. Όταν μιλάμε λοιπόν για ποιότητα, ταχύτητα και δυνατότητα, χωρητικότητα, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αρκετά καλοί στον ψηφιακό τομέα. Και να σας πω και το εξή. έχουμε τέλεια σενάρια για τον ποιο αριθμό αυτοκινήτων θα έχουμε στους δρόμους της Ευρώπης το 2030. Τι φορτία θα έχουμε. Η αύξηση των οδικών μεταφορών, σιδηροδρομικών μεταφορών, αεροπορικών μεταφορών είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε επακριβώς. Γνωρίζουμε όμως λίγα πράγματα για την ανάγκη μεταφοράς δεδομένων. Σας το λέω από τώρα, οι ποσότητες ε, ο όγκος των δεδομένων που θα μεταφέρονται θα ε, αυξάνεται εκρηκτικά με την βιομηχανία 4.0 με τον τομέα της πληροφορικής, με την άμεση επικοινωνία μηχανών μεταξύ τους, με το ίνερ, με τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Η ζήτηση για μεταφορά δεδομένων θα αυξηθεί εκθετικά. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο να πάμε από τα 3 στα 30 Mbps, ε, ούτε στα 100 δεν αρκεί. Μιλάμε για τα χίλια, Μιλάμε για ταχύτητες πάνω από τα 100 Mbps. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με τα δίκτυα των οπτικών ινών και την πέμπτη γενεά έτσι ώστε πανευρωπαϊκά να υπάρχει μια κάλυψη ψηφιακών υπηρεσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τώρα. Να σας πω κάτι άλλο για να γίνει πιο κατανοητό. Αν πάμε με τα αυτοκίνητα από τις Βρυξέλλες ε, στο Λουξεμβούργο, στο Ζαρμπρούκεν, Καζούι, Στουτγάρδη, Μόναχο για να φτάσω στο Σάλτσμπουργκ και το Λίντς μπορώ να πω ανα πάσα στιγμή που βρίσκομαι είτε στις Αρδένες είτε στις ε, στη Σουηδία ε, και άμα κινδυνεύω παίρνω ένα τηλέφωνο κτλ. Ε, αυτό έχουμε κάνει λοιπόν στα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν διόδια, δεν υπάρχουν ε, έλεγχος διαβατηρίων, τελωνία και λειτουργούν τα πράγματα πάρα πολύ απλά πηγαίνοντας από την χώρα στην ε, α στη χώρα β. Και αυτά χρειαζόμαστε. Τέταρτη, πέμπτη γενιά wireless ε, και βεβαίως ε, επένδυση στις οπτικές σύνες. Αυτά είναι ακόμη σημαντικότερα από την κατασκευή δρόμων και σιδηροδρόμων. Έχουμε ήδη το σχέδιο Juncker το οποίο συζητιέται και θα πρέπει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λαμβάνει το δυνατόν περισσότερα μέτρα για ευρυζωνικότητα, για συγχρηματοδότηση ψηφιακών ε, διόδων νομίζω πως είναι η σημαντικότερη πρόκληση που υπάρχει για τις ευρωπαϊκές υποδομές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προετοιμάζουμε και την οδηγία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια δεδομένων. Με, τους, ε, με τον συνάδελφο σας εδώ πέρα είχαμε πάει και μιλήσαμε σε ένα μεγάλο συνέδριο για την ψηφιακή ασφάλεια. Η βιομηχανία 4.0 κυρίες και κύριοι θα λειτουργήσει μόνο εάν ο πολίτης εμπιστεύεται το ψηφιακό νέφος και τις ψηφιακές υποδομές. Και γεγονός είναι πως και η βιομηχανική κατασκοπία του αύριο δεν θα λαμβάνει χώρα μέσα στο εργοστάσιο, με τη φωτογραφική μηχανή να ανοίξουμε τον ντουλάπι να βρούμε τα σχέδια. Θα γίνεται μέσω δεδομένων, μέσω των συστημάτων δεδομένων ναι ήδη σήμερα, ναι, ναι, βεβαίω εννοείται. Και αύριο και μεθαύριο, ναι. Λαμβάνει σήμερα, ναι, λαμβάνει σήμερα χώρα. Εγώ θέλω να το εμποδίσω αύριο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να βοηθήσετε να καταλήξει ε, κάπου αυτή η οδηγία. Μου φαίνεται πως ε, ήταν επιτυχημένη η λομπίστες των ε, OTTs γιατί θέλουν να συμπεριλάβουν και τις ε, πλατφόρμες. Χρειάζεται λοιπόν μια κουλτούρα επενδυτική και αυτό νομίζω πως μπορεί να αποτελέσει έναν κρίσιμο παράγοντα για την ε, οικονομική περιφέρεια που λέγεται Ευρώπη γιατί δεν είναι τόσο σημαντική ασφάλεια των δεδομένων σε άλλα μέρη του κόσμου. Επίσης έχουμε την οδηγία TIS η οποία νομίζω έχει συζητηθεί αρκετά και είναι σχεδόν αδιάφορο το τι θα προκύψει. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να λάβουμε μία απόφαση γιατί ε, αμέσως μετά την απόφαση θα πάμε στην μεταρρύθμιση, την ε, επόμενη μεταρρύθμιση του δικαίου του τηλεπικοινωνιακού στην Ευρώπη. Το χρόνο θα υποβάλουμε νέες προτάσεις για μια σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία στην Ευρώπη για ανταγωνισμό και επενδύσεις και για τις τηλεπικοινωνιακές μας επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα όπως το roaming, η ουδετερότητα του δικτύου και το φάσμα. Εγώ σας παρακαλώ ζητήστε από τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να μιλήσουν για συντονισμό συχνοτήτων οι καιροί των εθνικών δημοπρασιών έχουν περάσει. Όταν μιλάμε για πέμπτη γενιά, οι διαγωνισμοί δεν μπορούν παρά να είναι ευρωπαϊκοί. Για, την, ε, για το roaming συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει πλέον να περάσει στην ιστορία και μιλάμε για μεταβατική περίοδο. Είμαι σίγουρος πως σε ένα έως τρία χρόνια θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο χρέωσης κινητής τηλεφωνίας. Όταν ήμουν νέος υπήρχαν τοπικά και υπεραστικά τηλεφωνήματα και τώρα υπάρχουν εθνικά και διεθνή. Η εσωτερική αγορά χρειάζεται μία τηλεφωνική μονάδα. Γι' αυτό θεωρώ πως η περιαγωγή σε λίγο χρόνο θα ανήκει στην ιστορία και η ουδετερότητα του δικτύου τώρα. Πρέπει να αποφύγουμε κάθε είδους ε, διακριτική μεταχείριση για μικρούς και μεγάλους. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι χρειαζόμαστε προς το γενικό ε, συμφέρον, δηλαδή συστήματα παραδείγματο χάρη ε, της κυκλοφορίας ή της υγείας, ηλεκτρονικής υγείας. Εκεί δηλαδή όπου αποδεικνύει η τεχνολογία και η επιστήμη πως μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και χρειάζεται εγγυημένη ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων. Πρέπει να γίνει αυτό, αλλά μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, αποφασιστικό για εμένα είναι πέρα από την υποδομή, τις υποδομές και την ρύθμιση μια υπάρξη και ένα σύγχρονο τοπίο έρευνας. Έχουμε λάβει επαρκή κονδύλια για ερευνητικά έργα, με τη βιομηχανία, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Από το cloud computing μέχρι τα big data, από βιομηχανικά έργα του αύριο, όλες οι ερευνητικές δυνατότητες αυτές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Και εκεί πέρα υπάρχει ένας... υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και σκοπεύουμε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό copyright και να μεταρρυθμίσουμε βεβαίως ε, το θέμα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Τι εννοώ παραδείγματος χάρη, εάν η αυστριακή ραδιοτηλεόραση ή το RAI ή το BBC ή η γαλλική τηλεόραση ή το CDF προβάλλει κάτι στην τηλεόραση έχει απέναντι, έχουν απέναντι τους ε, υπηρεσίες όπως ε, ε, video on demand υπηρεσίες όπως το Netflix, το Amazon κτλ. Οπότε οι μεν πρέπει να προστατεύσουν τους νέους. Πρέπει να λάβουν υπόψη την, το κοινωνικό σύνολο, έχουν περιορισμούς στις διαφημίσεις και πάρα πολλά. Ενώ οι υπόλοιποι, οι πλατφόρμες δεν χρειάζεται να σέονται τίποτα και δεν υπεύθυνει για το περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού. Γι' αυτό εξετάζουμε το εάν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ε, της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα μπορούμε να εκδώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, να δημιουργήσουμε κάποιες ε, υποχρεώσεις για τους ε, OTTs, ανεξαρτήτως αν είναι στην Ευρώπη ή στην Καλιφόρνια όπου είναι συνήθως. Μετά, το θέμα της βιομηχανίας. Κυρίε και κύριοι, οι Αμερικάνοι, και εγώ αγαπώ την Αμερική, έχουν μια σαφή στρατηγική. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή υπεροχή για να δημιουργήσουν μια συνολική υπεροχή στην οικονομία. Δηλαδή η Google και η Apple θα περάσουν στην κατασκευή αυτοκινήτων, η Amazon θα καταλάβει τον χώρο του βιβλίου, το PayPal, τον χώρο των πληρωμών, θα είναι στο επίκεντρο των ασφαλίσεων επίσης και όποιος έχει τα δεδομένα θα έχει την δύναμη. Εσείς αγοράζετε ένα iPhone από την Apple και ε, αν δεν διαβάσετε τους ε, όρους, ε, πατήσατε συμφωνώ και πηγαίνετε από τις Βρυξέλλες ε, στη Στουτγκάρδη ε, με τα μάξι 4 η ώρα το πρωί και χιονίζει, ξέρει περισσότερα η Apple από ότι η General η ασφαλιστική σας εταιρεία. Ξέρει ότι οδηγάται επικίνδυνα και γρήγορα. Σε λίγα χρόνια λοιπόν θα μπορεί να σας αξιολογήσει πολύ καλύτερα από την ασφαλιστική εταιρεία. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για τη βιομηχανία, μιλάμε για το εμπόριο, την οικονομία, τη βιοτεχνία, την τραπεζική 4,0 όλα αυτά. Ολόκληρη πραγματική οικονομία λοιπόν. Γι' αυτό ε, κινδυνεύει η οικονομία μας πολύ περισσότερο από τους φόρους ή το εργατικό κόστος ή την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων. Χρειάζεται λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα μας δώσει περισσότερη ψηφιακή κυριαρχία, θα δημιουργήσει μία ενιαία και αγορά και μετά μαζί με την οικονομία μας, τις επιχειρήσεις μας θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά τα δεδομένα για να έχουμε σχέσεις με τον πελάτη, να αυξηθεί η ποιότητα, να βελτιωθούν οι διαδικασίες, όλα αυτά να περάσουν στην παραγωγή. Και είναι σαφές πως η αυτοκινητομηχανία είναι ο πρώτος κλάδος που θα επηρεαστεί, μετά η ε, κατασκευή εξειδικευμένων ε, μηχανημάτων και ακολουθούν οι υπόλοιποι κλάδοι. Οπότε η ψηφιακή αυτή ε, Ένωση, γιατί η ψηφιακή τεχνολογία είναι μόνο μια πλατφόρμα, αλλά η ψηφιακή ένωση επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, τη δημιουργία προσθέμενης αξίας, της ε, βιομηχανική ικανότητα. Είμαστε λοιπόν στο κέντρο όλων αυτών και σας παρακαλώ ως νομοθέτες, αλλά και ως ε, αρμόδιους για τον προϋπολογισμό, να σταθείτε στο πλευρό μας και θα ήθελα να σας ζητήσω πιο γρήγορη και αποτελεσματική νομοθεσία από ό,τι συνήθως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση που μας κάνατε για τα προβλήματα της ψηφιακής ενίας αγοράς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ήταν ε, μια άκρος πολιτική προσέγγιση στο θέμα και εμείς έχουμε ευθύνη ενώπιον των πολιτών μας για την πρόθεση του θέματος αυτό. Να περάσουμε λοιπόν στους ομιλητές από πλευράς ΕΛΚ, η κυρία Πιλάρ Τρικαστίγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα για άλλη μια φορά, μια τόσο σημαντική στιγμή προκειμένου να αντιληφθούμε τι σημαίνει ο στόχος και η πρόκληση μιας ε, ψηφιακής οικονομίας και μιας ε, ψηφιακής κοινωνίας θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής κοινωνίας είναι σαν ένα ε, τρένο υψηλής ταχύτητας χωρίς σταθμούς και η Ευρώπη δεν μπορεί να βρίσκεται στο τελευταίο βαγόνι ούτε καν στα μεσαία βαγόνια. Πρέπει να βρίσκεται στο ε, βαγόνι του μηχανοδηγού. Πρέπει να έχει τα ενία και αυτή είναι η ευθύνη μας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σαφές και το εξηγήσατε κι εσείς πάρα πολύ καλά, επομένως δεν θα επιμείνω εδώ για να μην σας καθυστερήσω. Η ενιαία αγορά είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ψηφιακή ένωση. Εντός όμως της ενιαίας αγοράς, η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της ενέας αγοράς, αυτής της κλίμακας που επιτρέπει στην ευρωπαϊκή οικονομία να είναι ανταγωνιστική υπό πολύ πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς και χρειάζονται όλες αυτές οι πτυχές τις οποίες αναφέρεται. Εγώ θα σταθώ μόνο σε δύο. Πρώτον, Βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, κατάστασης που μας επιτρέπει πολύ σύντομα να έχουμε μια ε, συμφωνία η οποία θα είναι υποφελής για όλες τις πλευρές και κυρίως για τους καταναλωτές, διότι περί αυτού πρόκειται για την περιαγωγή και την ε, ανοιχτή ουδετερότητα του δικτύου και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό το τελευταίο βήμα. Εδώ απευθύνομαι στην Επιτροπή μας, διότι θα γίνει και μια ενημέρωση σήμερα το απόγευμα και καταλαβαίνετε και πώς ε, θα σας περιγράψω πώς έχει κατάσταση και πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η τελευταία προσπάθεια και πρέπει να γίνει αυτές τις τελευταίες ημέρες. Και πραγματικά εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι έχουμε συνειδητοποιήσει την πρόκληση και τη δέσμευση και αυτό το πολιτικό και ηθικό καθήκον που έχουμε ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών που θα πρέπει να τους ε, ε, δώσουμε αποτελέσματα. Δεύτερον, Χρειαζόμαστε ηγεσία. Εγώ το γνωρίζω διότι είμαστε εδώ πάνω από 50 χρόνια. Γνωρίζω ότι εσείς είστε ένας πολύ αποφασιστικός πολιτικός που δεν διστάζεται ενώπιον των προβλημάτων και των προκλήσεων και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ε, και με τη βοήθεια του ε, Προειδοάνση, αλλά και μαζί σας που σας γνωρίζουμε τόσα πολλά χρόνια, να έχουμε πραγματικές ηγέτες στο τομέα. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ηγέτες, διότι τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα και η πολιτική χρόνια εν γέννη είναι πολύ αργή και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι πολύ πιο αργή. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατάλληλους ηγέτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει τα ενία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία έχει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να πιέσει το Συμβούλιο, αλλά ταυτόχρονα ε, πρέπει να έχει και αυτές τις πολύ σημαντικές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν απαραίτητη η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τίποτα. Τέλος, ε, κύριε Επίτροπε, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και είναι πολύ αργά τα πράγματα, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια δημιουργική προλητική προς αυτό ε, την κατεύθυνση με συγκεκριμένους προσανατολισμούς. Όσον αφορά την νομοθεσία, ε, υπάρχουν και προτάσεις που δεν αφορούν νομοθεσία ή που είναι πιο ήπια νομοθεσία και μπορούν να εφαρμοστούν ε, όπως ε, πολύ επέμεινε και ο συνάδελφος για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατάλληλες προτεραιότητες και να πάμε πραγματικά στην καρδιά του προβλήματος, να ξέρουμε περί τίνος θέλουμε να νομοθετήσουμε. Ιδάλλως θα είναι αδύνατο, θα φτάσουμε στο τέλος της θητείας και θα είμαστε λίγο καλύτερα από εκεί που ξεκινήσαμε, αλλά δεν θα έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ντανίκα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι, ότι είμαι πολύ χαρούμενος σας βλέπω εδώ. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Αναφερθήκατε σε κάποιες ιδέες που είχαμε διακούσει κατά την ακρόασή σας. Και χαίρομαι γι' αυτό. Ήρθε πια η ώρα η Ευρώπη να φτιάξει την ιστορία επιτυχία σε σχέση με την κινητή τηλεφωνία. Πριν από μερικέ δεκαετίε εμεί ήμασταν μπροστά. Και τώρα πρέπει να πείσουμε ότι είχαμε την πρωτοκαθεδρία και μπορούμε να τη διατηρήσουμε γιατί τη χάσαμε δυστυχώ με το 3G και το 4G. Τώρα έχουμε φτάσει στο 5G. Μία δυνατότητα για ανάκαμψη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερο τη σημασία αυτή τη ευκαιρία. Μπορούμε λοιπόν να διαθέσουμε τα κονδύλια που χρειάζονται για να προωθηθεί το 5G και να ολοκληρωθούν τα σχέδια. Πρέπει. Ξέρω ότι και στο σχέδιο Juncker υπάρχει αυτή η πρόταση. Το σχετικό κονδύλιο έχει διασωθεί ούτως πίν. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο λοιπόν φαίνεται να καταλήγουν σε μια κάποια συμφωνία για το στόχο και όπως είπα 5G, υποδομές, επενδύσεις στις υποδομές που είναι πολύ σημαντικές. Αλλά πώς θα γίνουν, πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι υποδομές και οι επενδύσεις. Όλα αυτά τα θέματα τα έχω υπογραμμίσει και στο παρελθόν. Η κυβερνοασφάλεια επίσης, ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, κέριο για οποιοδήποτε έργο θέλουμε να προωθήσουμε στην Ευρώπη. Ε, και πιστεύω ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα το οποίο να μας ε, εξασφαλίσει ένα είδος πιστοποίησης με έναν οργανισμό τρίτο ή ένα σώμα υπεύθυνο για την κυβερνοασφάλεια. Επί θέλει κανείς να ανατρέξει σε μια ε, διαγραμμική υπηρεσία, χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες Φελπίν, και επενδύσεις. Ε, με ζητήματα, οι οποίε όμω είναι εκτεθειμένες στην κυβερνοασφάλεια και μετά έρχεται ένα άλλο επενδυτή, για τον οποίο όμως δεν έχουμε στοιχεία διότι δεν υπάρχει το σχετικό σύστημα κυβερνοασφάλειας που να μας μιλήσει για την ε, διαβάθμιση, για την ε, αξιολόγηση του επενδυτή. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε λοιπόν. Και πρέπει να μπορέσουμε έτσι να λύσουμε και το πρόβλημα της ε, εμπιστοσύνης στην κυβερνοασφάλεια. Για να μπορεί ο πολίτης να αξιολογεί τις καταστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, Πρέπει να δείξουμε μια συνεπή στάση. Βέβαια, η Γενική Διεύθυνση για την ε, ψηφιακή οικονομία έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς αρμοδιοτήτων ε, συναφής. Αντίστοιχα αναπτύσσονται άλλες στρατηγικές και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα του ανατολισμού μας, της κατεύθυνσης προς την οποία κινούμαστε. Τη ψηφιακή λοιπόν, το ψηφιακό θεματολόγιο το διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, αλλά δεν έχει όλο το φάκελο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν ασυνέπειε, υπάρχουν προβλήματα και στις συνεννόηση ακόμα με τα κράτη-μέλη και τα διάφορα προσκόμματα. Το είδαμε αυτό άλλωστε και στο θέμα του, ε, της κινητής τηλεφωνίας, όπου είχε τοποθετηθεί η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, αλλά πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα και ε, γενική κάλυψη μηνύματα. Πρέπει να κοιτάξουμε τις τεχνολογίες του μέλλοντος επίσης. Γιατί μιλούμε για συστήματα ε, όπως το Raising the Volume, ε, πρέπει όμως να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι με μία φωνή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα εκ μέρους του ECR. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσία σας εδώ και την παρουσίασή σας. Είναι ο κύριος Κρόμπασης. Ε, χαίρομαι που είσαστε τόσο προσιλωμένος στην ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Έχω κάποια τεχνικά ζητήματα να ρωτήσω. Και τις ιδέες σας από τις υποδομές, σε σχέση με τις υποδομές. Ξέρετε, όταν περάσαμε από το αναλογικό στο ψηφιακό σύστημα, υπήρξαν κάποιες πρώτες λύσεις που μας έδιναν τις ψηφιακές ε, δυνατότητες ασύγκριτα καλύτερες από αυτό που είχαμε στο παρελθόν και έτσι το HDH ή το, τα ασυγχρονικά συστήματα το σύστημα των ATM μπόρεσαν να αναπτυχθούν. Τώρα μιλούμε για ασύρματη τεχνολογία και περαιτέρω βήματα τα οποία όμως φαίνεται να μην προχωρούν και αναφέρομαι σε προσκόμματα που προβάλλουν τα κράτη-μέλη ή που γνωρίζουν τα κράτη-μέλη λόγω διαφορετικών συστημάτων και ότι ο στόχος και η βάση είναι η ίδια. Χρειάζεται λοιπόν μια σειρά από ιδιαίτερες προσπάθειες να αναπτυχθεί σε σχέση με το δυναμικό του δικτύου, παραδείγματι. Και πρέπει να αλλάξουμε τεχνολογίες για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Σε μερικές περιπτώσεις ε, η λύση που προβλήθηκε ιδιαίτερα ήταν το fiber to desk, ε, οπτικές σύνες ε, ενσύρματη διασύνδεση. Αυτό όμως παρά μερίστηκε ως μη αποτελεσματικό. Μετά είχαμε το HTML που θεωρήθηκε ότι δεν ήταν επαρκές και θέλω να ρωτήσω το εξή. Όταν ε, αναλογίζεστε διαφορετικές επιλογές, εννοείται τελείως διαφορετικές λύσεις. Οπτικές είναι σε παραδείγματι. Είναι μια λύση την οποία επιδιώκεται ή κυρίως θέλει να κοιτάξετε το δυναμικό με χαλκό επί παραδείγματι. Γιατί αν θέλουμε πάνω από 100 MB δυναμικό θα είναι δύσκολο. Ξέρω ότι κάποιοι από τους παρόχους προσφέρουν τέτοιες λύσεις, όμως ε, συχνά δεν τηρούν τα υπεσχημένα λόγω των τεχνικών περιορισμών στη, στη μεταβίβαση των δεδομένων. Με τις επενδύσεις λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα ε, προβλήματα που επισημαίνω. Αλλά τι είδου επιλογές θα κάνει η Επιτροπή ως προς τις τεχνολογίες, τι είδου επενδύσεις θα προωθήσει και μια νομική ερώτηση για το μισητό αυτό πρόβλημα της περιαγωγής που τόσο πολύ μισάει ο πολίτης. Ξέρουμε ότι η λύση είναι στα χέρια κάποιων ε, κρατών μελών, η France Telecom, η Deutsche Telekom, ε, δεν έχουν συμφέρον να μειώσουν τα τέλη περιαγωγής, φοβούμενες ε, ότι θα χάσουν έτσι την επίδρασή τους στην αγορά. Πώς λοιπόν βλέπετε εσείς την κατάσταση αυτή και ίσως από τη θεώρηση της γερμανικής αγοράς πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τη δυνατότητα για ε, μείωση και εξάλληψη των ε, ε, τελών περιαγωγής χωρίς τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ για την παρουσίαση και συγχαρητήρια για τη στρατηγική σας, διότι καθορίζει σαφέστατα τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η ψηφιακή στρατηγική. Είναι μοχλός καινοτομία και άρσης φραγμών φυσικά και χωρίς να δημιουργήσουμε καινούριου. Ακούγοντα αυτά που μα είπατε σήμερα, πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Τελικαστήγιο Βέρα ότι χρειαζόμαστε ηγεσία. Δεν χρειάζεται να μιλούμε μόνο για του κινδύνου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και της ευκαιρίας που ε, μπορεί να προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά για τη βιομηχανία μας. Επειδή είμαστε Επιτροπή Βιομηχανίας, ε, ο βασική τομής ε, ε, Ενδιαφέροντό μας ε, σχετίζονται με αυτό. Πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε την ε, ψηφιακή οικονομία και πώς μπορούμε να έχουμε και ανάπτυξη. Αναφερθήκατε στη στρατηγική και ξέρω ότι η στρατηγική περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των διαδικτυακών στοιχείων και τις διάφορες πλατφόρμες που έχουμε. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς διαδικτυακή πλατφόρμα και πώς να την ορίσουμε, επομένως δεν ξέρουμε και τι προβλήματα υπάρχουν. Αναφέρατε και προηγουμένως ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος ρυθμιστικός φορέας ο οποίος θα υποπτεύει αυτές τις πλατφόρμες. Ε, πρόκειται απλώς για μία αξιολόγηση που θα γίνεται ή είναι ένα σχέδιο να υπάρχει ρύθμιση για αυτές. Θα μπορούσατε να με το σχολιάσετε λίγο πάνω. Όσον αφορά το copyright, τα πνευματικά δικαιώματα, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά για το ε, πολιτιστικό περιεχόμενο. Αυτό θέλουν οι καταναλωτές, ε, το να ε, αρνούμαστε να πληρώσουμε, ε, να πουλήσουμε, απλώς δημιουργεί παραπάνω πειρατεία. Επομένως, πότε θα υπάρχει μεταρρύθμιση για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το θέμα είναι πώς θα προχωρήσει η ολοκλήρωση. Αν υπήρχε νέα αγορά τηλεπικοινωνιών, θα μπορούσα ίσως να έχουμε αρκετές εταιρείες στην αγορά, μεγάλες εταιρείες και να υπάρχει ακόμα ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Πώς ε, προβλέπετε ότι θα εξελιχθούν αυτές οι αγορές. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ βεβαίως καταρχάς ότι έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι πρέπει, όπως είπατε κι εσείς, να μιλάμε όχι μόνο για ψηφιακή επανάσταση, αλλά και για βιομηχανία 4.0, όπως είπατε κι εσείς. Δεν υπάρχουν μόνο θέματα τεχνολογικά, αλλά θέματα και διοντολογικά. Πρέπει να κοιτάμε τον άνθρωπο. Ε, ισορροπία μεταξύ εσωτερική αγοράς και ε, βασικών δικαιωμάτων θεμελιωδών ελευθεριών. Μου φάνηκε ενδιαφέρον το παρα παράδειγμά σας θα πρέπει να δούμε ωστόσο τι είδους αποτελέσματα μπορούν να δώσουν ε, τα μάτια του δικτυού, ανάλογα με το αν θα είναι μικρά ή μεγάλα, δεν θα συζητήσουμε τόσο πολύ το μέγεθος όσο το αποτέλεσμα και πόσο μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα. Επίσης θα ήθελα ισορροπία, όπως έλεγα, μεταξύ εσωτερικής αγοράς και δικαιωμάτων των πολιτών. Κάποια αισθήματα επομένως πρέπει να τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Κατάργηση της περιαγωγής, ιδιαιτερότητα του δικτύου είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε γιατί από τις που βλέπουμε στο Συμβούλιο νομίζω ότι πηγαίνουν κάπως στη χάρπαστα. Υπάρχει ένα έγγραφο θέσεων για την ουδετερότητα του δικτύου από το Συμβούλιο, το οποίο φαίνεται να μην δίνει ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα ή να μην θέλει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Εσείς λοιπόν πώς μπορείτε να επηρεάσετε ιδιαίτερα τα κράτη αυτά ε, μέσα από τις συζητήσεις ε, ώστε να αλλάξουν θέση. Για τα τέλη περιαγωγής υπάρχουν σαφείς αποφάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θέλουμε να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής στην ουσία, όχι τυπικά μόνο και γι' αυτό πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε λύσεις. Το ίδιο για την ασφάλεια στη του διαδικτύου, Μεγάλε συστήσει και χτε ακόμα στην Ολομέλεια και παρούσα για την ασφάλεια. Αλλά το θέμα είναι τι είδου μέσα θα διαθέσουμε για να προχωρήσουμε στις λύσεις αυτές. Έρευνα, επιστημονική υποστήριξη. Τι είδους κονδύλια θα δώσουμε για να στηριχθούν αυτές οι επιλογές. Αυτά θέλουμε την γνώμη σας και επίσης ε, ε, για το θέμα του geoblogging. Αναφέρεται σαν να είναι κάτι το οποίο είναι αδικαιολόγητο και δεν πρέπει να υπάρχει και πρέπει να ε, μην γίνεται. Ναι, αλλά τι σημαίνει, σε τι είναι αδικαιολόγητο και πώς πρέπει να μην γίνεται. Θέλω πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τομέα, φορείς, ενώσεις που τα γνωρίζουν τα πράγματα στην πράξη έχουν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες και νομίζω θα πρέπει να τους εμπλέξουμε στη συζήτηση. Δεν πρέπει στο, στην ε, αναζήτηση λύσεων να θυσιάσουμε τα δικαιώματα του πολίτη, κάτι το οποίο πολύ συχνά έχει συμβεί. Πρέπει να αγωνιστούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να λησμονηθούν αυτό. Τίποτε δεν είναι αυτόνομο, δεν μπορούμε δηλαδή να επικεντρωθούμε μόνο σε ζητήματα βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογίας και να ξεχάσουμε τον πολίτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεωπρόεδρος. Οι λοιποί συνάδελφοι παρακαλώ να περιοριστούν στα δύο λεπτά. Έκαστος ο κύριος Παουλ Ρούμπιχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Το κοινοβούλιο με μεγάλη πλειονοψηφία η απεφάσισε ότι δεν επιτρέπονται οι επιβαρύνσεις για τέλος περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία και πρέπει να καταργηθούν. Εδώ βλέπουμε ότι παραμένουν ενώ έπρεπε να έχουν απαγορευτεί εφέτος το αργότερα μέχρι του χρόνου τα τέλη περιαγωγής. Και αυτό ήταν μια ε, ανεπιφύλακτη αποφάση του Κοινοβουλίου. Πάντως βλέπουμε ότι παραμένουν τα, τα τέλη αυτά από το ένα κράτος το οποίο μπορεί να κοστίζει μία μονάδα του gigabyte, παραδείγματι 2.30 στην Αυστρία σήμερα, μπορεί να εκατονταπλασιαστούν όταν πάμε σε ένα άλλο κράτος. 240 ευρώ μπορεί να μου κοστίσει εμένα το γιγαμπάιτ από την Αυστρία στη Γερμανία. Και μέχρι και 2004 ευρώ το gigabyte για κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως ε, ε, η οποία επιβάρυνση ή τέλος περιαγωγής για ορισμένα κράτη μπορεί να φτάσει και 19.000 για το gigabyte. Λοιπόν, πώς θα καταφέρω εγώ να ξέρω ότι έχω 2,4 στην Αυστρία, 240 στη Γερμανία, 2.040 στην, ή 4 στις κοντινές χώρες και μέχρι 19.000 στις λοιπές. Δεν είναι δυνατόν ο Ευρωπαίος πολίτης να ε, ε, γίνεται τέτοιο θύμα εκμετάλλευσης με το επιχείρημα ότι διαφορετικά δεν είναι δυνατές οι περαιτέρω επενδύσει κτλ. Πρέπει να έχουμε μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά. Το Συμβούλιο είναι πια καιρό να ακολουθήσει αυτές τις επιλογές, διότι διαφορετικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα ε, σημάνουν ότι θα χάσουν τη θέση τους στις αγορές μας οι πάροχοι της, ψηφια... της ε, κινητή στην ε, τεχνολογία, ώστε να θα μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί σε κάθε σημείο της Ευρώπης με ένα ενιαίο τιμολόγιο την ίδια τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις ξεκάθαρες δηλώσεις σας. Εγώ θα ήθελα η στρατηγική της ε, Κομισιόν να αναφερθεί περισσότερο στο θέμα τη βιομηχανία, τη βιομηχανία 4,0 και είναι θέμα πράγματι που επηρεάζει την ε, πραγματική οικονομία, τις τράπεζες, ασφάλειες, ε, όλο τον τομέα της ε, υγεία. Βλέπουμε ήδη πω ήδη επηρεάζεται η αυτοκίνητο βιομηχανία, οι μεγάλες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας επενδύουν σε Εταιρείε πληροφορικής γιατί χρειάζονται ακριβώς αυτή την ε, γρήγορη δικτύωση και οπωσδήποτε αυτό το θέμα θα είναι πολύ πιο σημαντικό στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε εδώ πέρα. Η ψηφιακή στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να δώσετε βάρος ακριβώς στην ε, πραγματική οικονομία και οπωσδήποτε ο παράγοντας του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η ΕΠΑ μας ε, έδειξε το, μας έδειξαν το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο επίπεδό τους. Η Ευρώπη είναι παγκόσμιος ε, ο πρώτος εξαγωγέας ε, ψηφιακών υπηρεσιών. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε περισσότερα Και σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπατε ότι θα μπορέσουν να δεσμευτούν κάποια ποσά ειδικά για αυτό τον ε, σκοπό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ακριβώς για να υπάρξει κάποια ψηφιακή επέκταση και ανάπτυξη. Δύο ερωτήσεις λοιπόν έχω να κάνω για το θέμα αυτό, τις οποίες ε, μπορείτε να απαντήσετε. Πρώτα απ' όλα για την χρήση των κονδυλίων, τι θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε, τι θεωρείτε πως μπορεί να γίνει με το ΕΦΣΕ το πακέτο αυτό. Γιούνκερ και δεύτερον την προηγούμενη φορά ο Επίτροπος Αντσίπη μας είπε στην Επιτροπή Ήτρε πως θα μπορούσε να υπάρξει κάποια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικό τομέα στη μονάδα η οποία είναι αρμόδια για την ψηφιακή ασφάλεια. αυτό το πράγμα και σήμερα γιατί είχαμε δει πως η Αμερικανική φορολογική ε, αρχή είδε, είχε, κάποια, είχε υποστεί κάποια επίθεση από Ρώσους hacker. Επίσης είδαμε χτες τι έγινε στο Βέλγιο, μείνανε χωρίς δεδομένα και χωρίς ρεύμα και άρα χωρίς ένα αέριο χώρο. Σας ευχαριστώ κυρία Κρέλ. Κύριε Επίτροπε, εκπλήσωμαι με αυτά που άκουσα γιατί πραγματικά συμφωνώ σε όλα μαζί σας κάτι το οποίο δεν μου συμβαίνει συχνά. Είμαι, δουλεύω στον τομέα της πληροφορικής, γι' αυτό γνωρίζω πόσο γρήγορα κινούνται αυτά τα συστήματα και πραγματικά χαιρετίζω το ότι δίνεται βάρος ε, στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Και θα χαιρόμουν πραγματικά κάποια θέματα που αφορούν την ψηφιακή ατζέντα να εγκριθούν κάπως πιο γρήγορα. Θεωρώ πως πρέπει επίσης να σκεφτούμε Μήπως ε, θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτη η νομοθεσία εκ των ε, προτέρων. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να, να θεωρούμε συνεχώς. Θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα και να είναι, όπως είπα, πιο ευέλικτο το σύστημα. Επίσης είμαι πεπισμένη πως ε, πρέπει να επιταχύνουμε όχι μόνο την νομοθεσία αλλά και τις υποδομές. Η Γερμανία λένε εντάξει είναι ανεπτυγμένη, τι ωραία, τι καλά, αλλά και για εμάς υπάρχουν κάποια ε, κενά ψηφιακά και όχι μόνο στην ύπαθρο αλλά και στις ε, πόλεις. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Ποια κίνητρα θέλει να δώσει Κομισιόν, εσείς δηλαδή, για να επιταχυνθεί η κατασκευή υποδομών με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το... Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι έχετε προβλέψει εδώ. Ευχαριστώ. Μαρτάν. Κύριε Μαρτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αν κατάλαβα καλά, δεν χρειάζεται μεγαλύτερη επιτελεσματικότητα στην Ευρώπη, διότι το να μας κατασκοπεύουν όλοι με πιο γρήγορες ε, ταχύτητες ε, ε, είναι επικίνδυνο. Εντάξει, ε, καλή κυβερνοασφάλεια, αλλά πρέπει να έχουμε και ασφάλεια για τους πολίτες μας. Τέλος πάντων, πέρα από τα αστεία, Υπάρχουν κάποιοι πυρογνώμονες που προβλέπουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη ε, για την επόμενη οκταετία επειδή δεν υπάρχουν και αυτό το είπατε κι εσείς ε, και είναι πολύ ε, ε, σημαντικό. Υπάρχει και η ψηφιακή ένδυα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Να αναφερόμαστε στους πολίτες που μπορεί να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή και στις νέες τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει να, να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους αυτούς που είναι αρκετά εκατομμύρια στην Ευρώπη και δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιστροφή στις επενδύσεις των ιδιωτών. Πώς μπορούμε να πείσουμε αυτούς τους ιδιώτες λοιπόν να επενδύσουν. Και επίσης ίσως χρειαζόμαστε και δημόσιες επενδύσεις. Και εδώ λίγο ξεκινάει και ένας φαύλος ε, κύκλος, διότι γνωρίζετε λίγο πώς έχει η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών των διαφόρων κρατών μελών τι μέσα μπορείτε να δώσετε ε, ώστε να υπάρξει όθηση για τις επενδύσεις. Επίσης, αναφέρεστε στην ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη, καλό αυτό, αλλά πώς μπορούμε να περάσουμε, τι ακολουθία ε, προβλέπετε ώστε από 28 εθνικές αγορές να περάσουμε σε μία ενιαία αγορά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπη. Ευχαριστώ η κυρία Μοντή. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω κι εγώ από αυτό. Θα σταθώ σε δύο τομείς. Ο ένας είναι υποδομές και χαίρομαι για την προσοχή που δίνεται στο θέμα αυτό. Υπάρχει ένα παράδειγμα στην περιοχή μου, ε, ένα πολύ γρήγορο ευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο ε, χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ευρωπαϊκά κονδύλια για να κατασκευάσει τις κατάλληλες υποδομές και να φτάσουν στους πολίτες. Και επίσης είναι πολύ εύκολο το εύστοχο το σχόλιο για ένα ψηφιακό κόσμο ο οποίος ε, διατίθεται ελεύθερα σε ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μας αλλά για ένα μεγάλο ποσοστό ε, υπάρχει αποκλεισμός και κυρίως στις περιοχές της Υπέθρου, που θα μπορούσαν να υπάρχουν και μεγάλα ωφέλη διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές ε, χαμηλόμιστες θέσεις εργασίας και επέκταση των υποδομών και στο ευρυζωνικό και στο φάσμα θα μας διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ίσως και πάλι αφορά τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στην οποία αναφερθήκατε. Χρησιμοποιώντας ίσως κάποιες από αυτές τις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πού υπήρχε καλή χρήση υποδομών και ανάπτυξης του ψηφιακού κόσμου, και να δημιουργήσει αυτέ τι καλή ποιότητα θέσει εργασία και ιδιαίτερα πριν φτιάξουμε τι θέσει εργασία χρειαζόμαστε και τι κατάλληλε δεξιότητε. Να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, νέους ανθρώπους, ε, πολίτες κατάλληλα εξοπλισμένους για να πληρώσουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε αυτή την αγορά που ελπίζουμε να εκμεταλλευτούμε και κάνουμε σε αρκετούς τομείς, όπως για παράδειγμα τις εφαρμογές. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την επιτυχία αυτή και να ε, χτίσουμε πάνω σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόιλ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ο συνήθω κύριε Επίτροπε ήταν πολύ επακριβής η ανάλυση στην οποία προβλήκατε των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών. Και βέβαια προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων. σε σχέση με την ταχύτητα, τους μεγάλους όγκους δεδομένων, την ευελιξία, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την ε, απορρίθμιση την οποία θέλουμε να ονομάσουμε ουδετερότητα του δικτύου, ε, δεν έχουμε κανένα περιθώριο και πρέπει και ευελιξία να πούμε ότι χρειαζόμαστε και ταχύτερα να προσφέρουμε τα δεδομένα και μεγαλύτερη να είναι των δεδομένων που ε, μπορεί να επεξεργαστεί το σύστημα αλλά θα ξεχάσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε μέσα σε μία μέρα. Νομίζω ότι πρέπει να συστήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο ειλικρινώς ότι όλα τα προβλήματα μέσα σε ένα πακέτο δεν μπορούμε να τα λύσουμε από την στην άλλη. Χρειάζονται μικρέ διορθώσει και το άλλο βέβαια ζήτημα είναι οι επενδύσει. Ναι, αλλά από πού θα βγουν τα λεφτά αυτά. Από το πακέτο Juncker. Καλή διασκέδαση. Ξέρω καν αν υπάρχει έτσι, αλλά και αν θα φτάσει και από πάνω. Πώς είναι δυνατόν να υποσχόμαστε στους ανθρώπους πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε. Γιατί μόνο αν υπάρχει ιδιωτικό χρήμα μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ιδιωτικό χρήμα τι σημαίνει να αναγνωρίσει ο ιδιώτης ότι αυτή η επένδυση με συμφέρει. Εκεί θα ρίξει τα χρήματά του. Αν όμω κάνουμε επιλογέ οι οποίε έχουν το συνέπειο ότι δεν θα μπορεί από την επένδυση να κερδίσει χρήματα, δεν θα γίνει επένδυση. Αυτό λοιπόν ο οποίο έχει ιδιωτικό κεφάλαιο στα πρέπει να θέλει και να επενδύσει. Εμείς πώς θα τα καταφέρουμε λοιπόν και έχουμε το θάρρος να τα καταφέρουμε. Σαλίνη παρακαλώ. Ο κύριος Σαλίνη βέβαια. Ε, όχι και μαντάμ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ καταρχάς για τον ενθουσιασμό σας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, διότι νομίζω ότι το πρώτο θέμα προκειμένου να ε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι σε θέση να ξεκινήσει με το απαραίτητο στένος είναι να υπάρχει πεποίθηση και ε, ε, κυριαρχία από πλευράς μας. Ελπίζω λοιπόν ο ενθουσιασμός σας να μεταλαμπαδεύετε και στους συναδέλφους σας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό κύριε Επίτροπε. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων σε θέματα ψηφιακού θεμετολογίου. Εγώ ασχολούμαι με την παλιού τύπου βιομηχανία. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι υπάρχει ανάγκη ε, μέσω όσμωσης να ε, περάσει και η ψηφιακή πρόκληση στη βιομηχανία η γεωργία. Εγώ προέρχομαι άλλωστε από την Ιταλία, μια χώρα που εκτός από βιομηχανική είναι και γεωργική χώρα. Οι νέες τεχνικές ε, ίδρευσης εκμεταλλεύονται τη χρήση δορυφόρων και μέσω αυτών οι ε, γεωργοί ε, μέσω του smartphone τους ξέρουν αν έχει αρκετό νερό σε μια περιοχή ή όχι. Λοιπόν, θέλουμε να την αναλάβουμε αυτή την πρόκληση και ελπίζω να την αναλάβουμε μέχρι τέλους. Και μια τάκα τώρα να σας πω. Ποιος είναι ο εχθρός αυτών των επενδύσεων. Η υπερβολική νομοθεσία, η υπερβολική ρύθμιση. Εμείς πριν αποκτήσουμε καλή νομοθεσία, χρειαζόμαστε λιγότερη νομοθεσία. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα μικρό βήμα προς τα πίσω και πρέπει εμεί να αποφασίσουμε ω μεγάλε χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεχόμαστε αυτό το κίνδυνο. Και όπως είναι γνωστό, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομοθεσία και δεν πρέπει να υπάρχει κρότ, ε, ε, κράτος, αλλά κάποιος που είναι αδύνατος κινείται καλύτερα από κάποιον που είναι παχύσερκος. Επομένως, το κράτος πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να έχει αθλητικό σώμα και αυτό είναι το ουσιαστικό. Επομένως, από αυτή την άποψη και με αυτό ολοκληρώνω, η σημασία ε, για μένα έγκυται στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ επενδυτή και πολιτικής. Ο επενδυτής όπως ακούστηκε σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς δεν πάει εκεί που υπάρχουν εγγύησεις. Ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος δέχεται περισσότερο από όλους τον κίνδυνο. Το μόνο το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ο επενδυτής είναι η γραφειοκρατία και οι υπερβολικές ρυθμίσεις. Για την περιαγωγή ακούστηκαν πολλά, για τις τηλεπικοινωνίες δεν επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλίνη. Ε, ζητώ συγγνώμη αλλά... Ε, θα προσέχω από εδώ και πέρα. Κύριε Μπόνη, ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον Επίτροπο για το πάθος και τον ενθουσιασμό του. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία για την επιτυχία μας. Καταρχάς καλή ηγεσία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ευέλικτη νομοθεσία. Συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε ευέλικτη νομοθεσία και επίσης λύσεις μη νομοθετικού χαρακτήρα όταν αναφερόμαστε στην εφαρμογή της ενέας ψηφιακής αγοράς. Τρίτον, επενδύσεις σε υποδομές. Αυτό είναι ουσιαστικό ζήτημα για το μέλλον και το τέταρτο είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης ε, της βιομηχανίας. Νομίζω ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιγράφει ε, πλήρως αυτή την οικονομία 4.0 όπως την ε, περιγράφεται. Ε, πρέπει να υπάρχουν νέοι στόχοι για την περαιτέρω συνεργασία μας και αυτό ε, είναι μια πρόκληση για σας ως Επίτροπο. Ε, ο κύριος... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για τα όσα μας είπατε με πολύ πάθος για την ψηφιακή εσωτερική αγορά και όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν και πολλοί συνάδελφοι μπορούμε νομίζω να προσυπογράψουμε όλα όσα λέτε και πραγματικά θα είναι θετικό να υλοποιηθούν αυτά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και αν γίνουν όντως θα πρέπει να σας δώσουν ένα ψηφιακό νόμπελ αλλά θα είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί όταν κανείς έχει ένα σχέδιο πρέπει να έχει και προτεραιότητες, πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητες. Ποιες είναι λοιπόν οι δικές σας προσωπικές προτεραιότητες που θέλετε όντως να υλοποιηθούν τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτά τα οποία παρουσιάσατε ως σχέδιο είναι κάπως πιο μακροπρόθεσμα. Ο ψηφιακό κόσμος θέλει να γίνονται όλα πιο γρήγορα, αλλά με βάση τα δεδομένα τη Ευρωπαϊκή πολιτικής θα αργήσουν λίγο αυτά. Εσείς προσωπικά τι θέλετε να δείτε τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δεύτερο ερώτημα. Οι συνάδελφοι το είπαν όλοι πως πριν μιλήσουμε για μια ψηφιακή επανάσταση πρέπει να επενδύσεις τις υποδομές. να τελειώνω. Είστε τώρα στην Κομισιόν προγραμματίσατε κι εσείς μαζί το πακέτο αυτό Γιούγκερ. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα ποσά και αν όντως θα πάνε αυτά τα ποσά για επενδύσεις στην ε, βριζονικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, μετά από την ε, συναρπαστική και επαγγελματική αυτή συζήτηση έχετε τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, το ερώτημα είναι πόσο χρόνο θέλουμε να ακούσουμε τους ειδικού, τους επιστήμονες, τους εμπειρογνώμονες και να είμαστε γρήγοροι παρόλα αυτά. Κοιτάξτε. Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων τον επεξεργάστηκε η κυρία Ρέντιν πριν από 2,5 χρόνια ε, και τον επεξεργάστηκε η και μπλοκαρίστηκε δύο χρόνια από το Συμβούλιο. Χωρίς κάποιο ε, λόγο. Οπότε σας παρακαλώ να δώσετε γρήγορα έντολη και γρήγορες διαβουλεύσεις μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Δεύτερο παράδειγμα. Όταν έχουμε τρεις συνεδριάσεις του Συμβουλίου το χρόνο για να περάσουν κατεπηγόντως νόμοι. Και εγώ ήμουν τον Νοέμβριο την τελευταία φορά στο Συμβούλιο στη συζήτηση αυτή και μετά τον Απρίλιο ε, έχουν φύγει έξι κυβερνήσεις. Έχουμε έξι νέους υπουργούς, Από τους 22 δε 18 στέλνουν κάποιον υφυπουργό ή γενικό γραμματέα, δεν στέλνουν καν υπουργό και ο οποίος είναι ένας υπάλληλος και μας διαβάζει ε, αυτά που του έχουν γράψει οι υπουργοί κάθονται και δεν ε, κοιτάνε και δεν λένε τίποτα και απλά κοιτάνε. Δεν, δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Είναι κάποιε ιεροτελεστίες. Ναι, να τα εξετάσουμε ει βάθο αλλά αυτό δεν αποκλείει το να κινηθούμε γρήγορα. Η οδηγία για τα οπτικοακουστικά είναι από το 2007 και τώρα αναθεωρείται. Εξετάζουμε τι αποδείχθηκε σωστό, τι ήταν λάθος, τι πρέπει να εξυγχρονιστεί, τι πρέπει να προσθεθεί. Και στο δεύτερο τρίμηνο του επομένου έτους ε, θα φέρουμε πιθανότατα μια νομοθετική πρόταση. Ε, δεν χρειάζεται να χάσουμε πια πάλι τόσο πολύ χρόνο. Γιατί σε αυτά τα τρία χρόνια εμφανίστηκε το Netflix, το Amazon, οι υπηρεσίες streaming, video on demand ε, έχουν εμφανιστεί μάλλον και θα αλλάξουν ξανά Οπότε πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο επίκαιροι. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει οι ή οι υπουργοί, ε, οι αρμόδιοι της να μπουν σε μία αίθουσα, να τους κλείσουμε και να μην βγουν μέχρι να βγάλουν αποτέλεσμα. Αν μπορεί δηλαδή να γίνει για την εκλογή του Πάπα, πρέπει να μπορεί να γίνει και στις δημοκρατίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει τσαπατσούλικα σωστά αλλά γρήγορα. Έτσι ώστε τελικά να βγει για τον ψηφιακό τομέα κάτι το οποίο θα πείσει τους πάντες ότι σε αυτόν τον τομέα κινούμαστε πιο γρήγορα, χωρίς διακοπές, με όλους τους εμπλεκομένους και όχι μόνο με τους πρέσβεις στην Κορεπέρ. Και αυτό πραγματικά μας ωφελεί να έχουμε κύρος στον ψηφιακό κόσμο, στον κλάδο εντός και εκτός Ευρώπης. Ουδετερότητα του δικτύου και roaming το ανέφεραν κάποιοι. Ε, σας ευχαριστώ. Έχετε έξυπνους ε, εισηγητές εδώ πέρα τις επόμενες εβδομάδες θα εργαστούν εντατικά και είχαμε και ένα πρόγευμα εργασίας, έχουμε ένα πρόγευμα εργασίας στο Συμβούλιο σε δύο εβδομάδες και στόχος είναι να λάβουμε μια απόφαση επί Προεδρίας. Το Λουξεμβούργο είναι προετοιμασμένο να συνεχίσει, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τον χρόνο που έχουμε ακόμα τον Ιούνιο για την ουδετερότητα του δικτύου. Θεωρώ πως το βάρος της αποδείξεως ε, πρέπει να μετατοπιστεί. Πρέπει οι υπηρεσίε υγείας, η ιατρική να αποδείξει τον ισχυρισμό πως η e-health, η ηλεκτρονική υγεία είναι δυνατή μόνο με χρόνο υστέρησης μιλισεκόντ. Και να υπάρχει έτσι ανοιχτή πρόσβαση του καθενός στην ψηφιακή υποδομή. Επίσης, ο τομέας των συγκοινωνιών πρέπει να αποδείξει το πού και το εάν υπηρεσίες ε, τέτοιες ε, είτε μιλάμε για υπηρεσίες ασφαλείας ή και αυτόματη οδήγηση είναι κάτι το οποίο ε, απαιτείται και τότε θα έχουν προβάδισμα προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και της οδικής ασφάλειας. Χωρίς όμως αυτό δεν θα γίνει τίποτα. Για να υπάρξει λοιπόν κάποιο προβάδισμα για ειδικέ υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι ισχύει κάτι τέτοιο. για να συμπληρώσουμε, όπως είπα, την ουδετερότητα του δικτύου με κάτι επιπλέον. Τώρα για το θέμα ψηφιακή ασφαλεία. Υπάρχει πέρα από την νομοθεσία και η, το θέμα των διαφόρων μικροπλατφορμών και των ΣΔΙΤ και για περαιτέρω εσωτερική ανάπτυξη τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην Κομισιόν, αλλά και για τον εξωτερικό κόσμο, στο Digit και στο Connect. Να φτιάξουμε κάποιες ομάδες εργασίας έτσι ώστε να κινηθούμε πιο γρήγορα από ό,τι το κάνουμε μέχρι στιγμής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε hacking, επιθέσεις στα δίκτυά μας και να βγάλουμε μετά και τα συμπεράσματα μας. Όταν έχουμε παραδείγματο χάρη αποδεδειγμένες επιθέσεις ε, που προέρχονται εκτός Ευρώπης ε, στα συστήματα τα δικά μας ε, και πιθανώ και επιθέσεις στην ψηφιακή υποδομή μυστικών υπηρεσιών που είναι εντό τη ευρωπαϊκή Ένωσης. Όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ψηφιακή ευαισθησία στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ε, υπόθηκε πως ε, στην ανακοίνωση που βγάλαμε για το DSM δεν ε, αναφέραμε αρκετά την βιομηχανική πολιτική. Μπορεί, αλλά συγκρίνεται την δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τα οχήματα και την κινητικότητα, αλλά η έρευνα για το αυτοκίνητο του αύριο είναι κάτι άλλο. Η εσωτερική ψηφιακή αγορά είναι μια βάση για ψηφιακή ε, πολιτική και πολιτική βιομηχανία. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή υποδομές, κανόνες, ε, προστασία των δεδομένων, ασφάλεια των δεδομένων είναι βάση αυτά βιομηχανικής πολιτικής. Η δικτύωση ε, και για την δικτύωση της ψηφιακής οικονομίας και της πραγματικής οικονομίας. Οπότε η ψηφιακή ένωση είναι το όραμα και η ψηφιακή ιστορική αγορά είναι το η αναγκαία αλλά όχι η ικανή συνθήκη. Με την, το 5G, την πέμπτη γενιά της ασύρματης επικοινωνίας του μέλλοντος έχουμε μείνει πίσω. Δώσαμε 750 εκατομμύρια ευρώ σε μια κοινοπραξία με τον κλάδο την βιομηχανία. Ο κλάδος δεσμεύτηκε να επενδύσει τα πενταπλάσια και μπορώ να σας πω πώς ε, πλησιάζουμε του υπόλοιπου Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Και στόχος πρέπει να είναι η Ευρώπη να μπει ταυτόχρονα στο, στην πέμπτη γενιά τη τηλεφωνία μαζί με Νότια Κορέα και Ιαπωνία, κάποια στιγμή το 2020. Ένα συναρπαστικό ερώτημα ήταν το θέμα των επενδύσεων στην ψηφιακή υποδομή. Κυρίε και κύριοι, χρειαζόμαστε νομίζω μια κατανομή των αρμοδιοτήτων. Ποιο είναι υπεύθυνο γιατί πράγμα και ποιο είναι ο στόχο. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει έχουμε ξεκάθαρε αρμοδιότητες στους δρόμους. Ποιοι είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι εθνικέ οδοί περιφερειακοί δρόμοι και δρόμοι αρμοδιότητος, αρμοδιότητος δήμων. Τα νοσοκομεία, στα σχολεία, είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Τι κάνει ο Δήμος, η περιφέρεια, το κράτος. Αντιθέτως, στην ψηφιακή υποδομή, στην ευρυζωνικότητα, υπάρχει χάος στις αρμοδιότητες. Και πρέπει τώρα να αποφασίσουμε στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker πώς έχει η κατάσταση στα κράτη-μέλη για να συγχρηματοδοτήσουν από τους προϋπολογισμούς, τι γίνεται με τις περιφέρειες, τι είναι αποδεκτό ως επιδότηση, τι γίνεται με τους Δήμους και τι βεβαίως είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν τα διαφορετικά προγράμματα που αυτή τη στιγμή ε, δεν χρησιμοποιούνται πάρα πολύ για ψηφιακή συγχρηματοδότηση και εγώ θα έλεγα πως ε, πολύ σημαντικότερο από τις ε, παρακαμπτήριες οδούς και τις μαρίνες είναι αυτό το πράγμα, η ψηφιακή υποδομή και το ΕΦΣΙ τις επόμενες μέρες θα αποφασίσουμε για τα κριτήρια του ΕΦΣΙ, τι θα συγχρηματοδώσουμε, πού μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο και να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και για την υπεθρό. Γιατί χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια μια πανευρωπαϊκή υποδομή όχι μόνο στις Μητροπόλεις της Ευρώπης αλλά και στις αραιοκατοικημένες περιοχές γιατί τα σχολεία χωρίς ψηφιακά μέσα ή το θέμα της ψηφιακής υγείας ή το θέμα της αυτόματης ε, οδήγησης έχει μόνο νόημα εάν δεν υπάρχουν κενά στην κάλυψη και όλη η Ευρώπη έχει πλήρη κάλυψη σε ταχύτητα και συμπεριλαμβάνω εδώ πέρα και την Ουκρανία, Δυτικά Βαλκάνια, Ελβετία και τα λοιπά σε αυτές τις υποδομές. Και μετά έχουμε το θέμα των κριτηρίων επιδότησης. Θα πρέπει να είμαστε νομίζω τεχνολογικά ουδέτεροι αλλά να έχουμε κάποια ποιότητα κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Τώρα αν θα είναι vectoring ή οπτικές ίνες ή ασύρματη τεχνολογία, αυτό θα το αφήσουμε ε, ή στα κράτη-μέλη ή στον ε, κλάδο. Εγώ τώρα... Δεν, ε, δεν μας είναι βέβαιος αδιάφορο αν μιλάμε για 3 Mbps ή 15 Mbps. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για το τι θα ενισχυθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η κυρία Κάλλας ε, με ρώτησε για τις πλατφόρμες. Αυτή μία έχουμε την περίπτωση του Google, από το οποίο θα, βγάλουμε, θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες ήταν οι εμπειρίες μας, ποιες ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές και το τι πρέπει να γίνει κατά της διακριτικής μεταχείρισης για ε, την ευθύνη για το περιεχόμενο και μετά θα αναλύσουμε την αγορά μας στο τέλος ε, του έτους για να γίνει μια πρόταση το εάν και σε ποιο βαθμό παράλληλα με τις ρυθμίσεις στα που έχουμε για τις λεπικοινωνιακές εταιρείες, για τις ραδιοτηλεοράσεις, θα κάνουμε και κάτι για τους, ε, ό, τις, τις ε, αυτές για τη μη διακριτική μεταχείριση, τις διαφημίσεις, ε, φορολογική μεταχείριση κτλ. Θεωρώ δε πως ε, η συγκέντρωση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών πρέπει να προσφέρει όχι λιγότερο αλλά καλύτερο ανταγωνισμό. Δεν μιλάμε για μονοπολία, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 200 ε, τηλεπικοινωνιακές εταιρείε οι οποίες δρούν κατά κανόνα μόνο στο κράτος μέλος τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, δώσουμε δυνατότητες για περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου. Εγώ προτιμάω 10 Ευρωπαίους που μπορούν να ανταγωνιστούν αντί για 300 που ο καθένας έχει την ε, γωνία του. Αναφέρθηκαν ερωτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πολύ σωστά. Έχω και με τη Βέρντι στην πατρίδα μου αλλά και με άλλες συνδικαλιστικά σωματεία ε, επαφές για να δούμε πώς μπορούμε να καταγράψουμε και τα πλεονεκτήματα σχέση με τον άνθρωπο, φερειπίν ε, ε, εργασία από το σπίτι, αλλά και τους κινδύνους σχετικούς με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βέβαια τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί ο τρόπος εργασίας στην βιομηχανία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η ψηφιακή επανάσταση να αποβεί εις του ανθρώπου, των εργαζομένων ανδρών και γυναικών και να μειώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο ή να εξαλείψουμε τελείως τα μειονεκτήματα. Ψηφιακή ευαισθησία. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε απόλυτη σωματική ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σε μια βιομηχανική μονάδα, στην πρέσα, στο, στην αλυσίδα παραγωγής του εργαζομένου, το ίδιο πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε και στον ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό καλούμε και τα επιχειρησιακά συμβούλια και γενικά τους φορείς του κλάδου να συμμετάσχουν και να δώσουν τις θέσεις τους για τα έργα που ε, σχεδιάζονται σε επίπεδο και να συμβάλλουν με τις ιδέες τους. Το geo-blocking, τελευταίο θέμα για σήμερα, ε, μεταφεροσιμότητα, ε, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με βάση λειτουργίας μιας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ένα κράτος το σημείο προσέγγισης. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι κατ' εξαίρεση μπορεί να είναι ένα κράτος το σημείο προσέγγισης. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή τρία, όπου δημόσιοι κρατικοί οργανισμοί τηλεοπτικοί ε, χρηματοδοτούνται μέσω τελών από τους πολίτες και έχουν την υποχρέωση της βασικής υπηρεσίας μέσα στα κράτη αυτά, όχι εκτός. Τα δε τέλη θα ήταν πολύ λιγότερο ευχερές να αιτιολογηθούν εάν από τη μία μέρα στην άλλη καταργούσαμε την έννοια της εδαφικότητας, δηλαδή τον περιορισμό στο εθνικό, στην εθνική επικράτεια. Δεύτερο, ε, τηλεοπτική διαφήμιση στον αθλητισμό, στο αθλητισμός και αθλητικές ε, ενώσεις, ε, στο ποδόσφαιρο λοιπά μας μιλούν για τη δυνατότητα να περιοριστεί ή όχι αυτή η έννοια της εδαφικότητας με το εξής επιχείρημα. Εάν παίζει το Αμβούργο κατά της άλλης τοπικής ομάδας του Αμβούργου του Σανκ τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει να μεταδοθεί σε μια άλλη χώρα. Γιατί δεν πρέπει να μιλούμε για κατάρριξη εδαφικότητας μόνο σε μία, ε, μόνο για τις μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου που έχουν το κύριο ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά για τις μικρότερες, τις πιο τοπικές και τα άλλα αθλήματα που δεν είναι τόσο δημοφιλή. Τότε μόνο πρέπει να δούμε την εδαφικότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ε, επηρεαστούν και οι αθλητικές ενώσεις. Θα έχω αντατικέ συνομιλίες μαζί τους επόμενες ε, εβδομάδες και μήνες και η Επιτροπή ε, Πολιτισμού και η Επιτροπή Βιομηχανίας θα πρέπει να εμπλακούν ασφαλώς αυτό και βέβαια πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για τον αθλητισμό για την κινηματογραφική παραγωγή και τις κινηματογραφικές ταινίες, οπωσδήποτε χρειάζεται μια διαφορετική λύση, γιατί δεν είναι δυνατόν η ευρωπαϊκή ε, κινηματογραφική παραγωγή να αντισταθεί διαφορετικά στην ε, ε, συντριπτική ανταγωνιστική θέση του Hollywood, του Netflix και της Google. Χρειάζεται λοιπόν να τηρηθεί μια αρχή εδαφικότητας τουλάχιστον σταδιακά ή προς το παρόν ένας ε, παραγωγός, ε, παραδείγματι, που θέλει να φτιάξει μια ταινία στην Αυστρία, θα πάρει ενίσχυση από την Αυστρία, ενδεχομένως να μπορέσει να προβληθεί και στη Γερμανία το πολύ. Μην ξεχνάμε ότι, έχουμε μόνο, ότι δεν έχουμε μόνο μία γλώσσα, έχουμε 24 διαφορετικές γλώσσες, δεν έχουμε μόνο μία ιστορία, έχουμε 28 διαφορετικές ιστορίες, συμφέροντα διαφορετικά, ε, ιδέες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μορφοποιούμε κάποιες προσωπικότητες. Ενδιαφέρον για να δει κανείς ε, στην Πορτογαλία, Φερρυπίν, μια γερμανική ταινία, 0,0%. Τίποτε περισσότερο. Ελάχιστε είναι αυτέ τι ταινίε οι οποίε έχουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να εξωτερώσουμε το, την πολιτισμική μα παραγωγή και πάνω από όλη την πολιτισμική πολιτιστική μα ιστορία, δεν είναι δυνατόν από τη μια μέρα στην άλλη να να ανοίξουμε τα σύνορα της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη για τον κινηματογράφο. Το geo-blocking έχει κάποια αξία λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα βέβαια της μεταφοράς. Πρέπει, αν είναι μια μεγάλη, ένας μεγάλος αγώνας ε, που παίζεται στην Αυστρία, να μπορώ να τον δω κι εγώ στην, ε, στις Βρυξέλλες εδώ γιατί με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε μικρός αγώνας και οποιαδήποτε αθλητική αναμέτρηση, αναμέτρηση ή μικρότερης εμβέλειας ε, πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραγωγή θα ε, κυκλοφορούν παντού στην Ευρώπη χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστώ πολύ τον Πέτρο Λεοπρόεδρο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε πάντα διαθέσιμοι να σας συναντήσουμε. Μας ενδιαφέρουν και χρειαζόμαστε συζητήσεις τέτοιες για την ψηφιακή οικονομία, για την συνεργασία μας. Δε. Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ καλή τα τελευταία έξι χρόνια. Δεν την ανακαλύψαμε πέρσι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, να περάσουμε τώρα στι συνεδρίες των συντονιστών και επιτρέψτε μου να ζητήσω από όσους δεν